Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρηματοδοτικής Βοήθειας. Καλώς ήρθατε κύριε Αντιπρόεδρε Νταμπρόμφσκης και κύριε Επίτροπη Μοσκοβισή. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Πριν από δύο εβδομάδες κάναμε την αποστολή μας στην Αθήνα, μια διερευνητική αποστολή που ήταν πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερα επιτυχής. Δεν θα σας κάνω τώρα την παρουσίαση του έργου της αποστολής, αλλά φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει τα σχετικά έγγραφα. Η αξιολόγηση προχωρεί προς θετικό συμπέρασμα με κάποια θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Αλλά οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται στο ίδιο μήκο κύματο. Υπάρχουν ε, κάποιες απόψεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημοσιονομικό κενό και δόθηκαν σημαντικές δεσμεύσεις και από τους θεσμούς και από την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Και τώρα περιμένουμε να ακούσουμε από τους δύο επιτρόπους τι έχουν να μας πούν. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι επί τη βάση των όσων είδαμε εμείς στην αποστολή, Νομίζω ότι θα έχουμε ένα θετικό συμπέρασμα όσον αφορά το Staff Level Agreement, τη Συμφωνία για το Επίπεδο Υπηρεσιών. Και νομίζω ότι ε, η συμμετοχή και μη ευρωπαϊκών θεσμών θα δυσκολεύσει την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης. Ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η αναθεώρηση για την Συμφωνία Επέδου Υπηρεσιών πριν από την Ερηνή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να μπορέσουμε να έχουμε και την τελική ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Δεν θέλω να βάλω κάποια προθεσμία, κάποια τελική προθεσμία. Σύντομα ήθελα να πω. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε από τον κύριο Ντομπρόφσκης και τον κύριο Μοσκοβισή τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές που υπάρχουν για την αναθεώρηση. Θα δώσω το λόγο στον Βάλτης Ντομπρόφσκης πρώτα και στη συνέχεια στον Πιέ Μοσκοβισή και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και απαντήσεις. Βάλτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα με αυτή την ευσυσταθήσα ομάδα εργασίας χρηματοδοτικής βοήθειας. Όπως είπε ο ίδιο ο κ. Γκουαλτιέρη, πρόσφατα έγινε μια διερευνητική αποστολή στην Αθήνα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για την εξέλιξη των εργασιών. Όπως γνωρίζετε, διεξάγονται ιδιαίτερα εντατικές διαπραγματεύσεις ε, και τώρα που μιλάμε και οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του περασμένου καλοκαιριού. Οι συζητήσεις στρέφονται γύρω από τα μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών ε, στόχων, ε, πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% μέχρι το 2018, μεταρρύθμιση των συντάξεων, ε, στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ανεξάρτητη αρχή εσόδων, νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, άνοιγμα των αγορών αερίου και ενέργειας και άλλα θέματα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν, αλλά βέβαια η πρόοδος εξαρτάται από τις ελληνικές αρχές. Αξίζει να τονίσουμε ότι τα πρόσφατα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί περισσότερο ανθεκτική από ό,τι αναμένεται πέρυσι το καλοκαίρι. Τα μακροοικονομικά δεδομένα που θα επικαιροποιηθούν και αρχές Μαΐου δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη προχωρεί καλά και ότι προχωρούμε προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ε, εάν η αναθεώρηση ολοκληρωθεί επιτυχώς τώρα και οι μεταρρυθμίσεις υλοποιηθούν εγκαίρως και με επιτυχία, η Ελλάδα μπορεί να αρχίσει να ανακάμπτει ήδη από το δεύτερο εξάμεινο του 2016. Από το περασμένο καλοκαίρι σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά για να υλοποιήσει την φιλόδοξη και μπροστοβαρή στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Τηρήθηκαν τα προαπαιτούμενα, δύο ομάδες προαπαιτούμενων, ε, ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε γιατί η Ελλάδα ακόμη πρέπει να υιοθετήσει σημαντική δέσμη μέτρων. Η Επιτροπή βοηθάει ενεργά την Ελλάδα με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Πέρυσι τον Οκτώβριο συμφωνήσαμε με τι ελληνικέ αρχέ ε, επί ενό σχεδίου τεχνική συνεργασία για την υποστήριξη διαφορετικών μεταρρυθμίσεων σε ε, τομεί προτεραιότητα όπω είναι η διοίκηση εσόδων, η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση τη διαφθορά, ε, τα ε, η, φραγμή, η ρυθμιστική φραγμή στον ανταγωνισμό, ιδιωτικοποίηση, δημόσιες συμβάσεις και μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Η τεχνική βοήθεια προσφέρεται από την Επιτροπή Απευθείας, καθώς και μέσω συμφωνιών με τα κράτη-μέλη και με διεθνείς οργανισμούς και συντονίζεται από την ε, Υπηρεσία Υποστήριξης Διαθετικών Μεταρρυθμίσεων που έχουμε ως Επιτροπή. Θα ήθελα όμως να είμαι σαφή ότι η Επιτροπή δίδει και συντονίζει την υποστηρικτική αυτή βοήθεια. Οι ελληνικές αρχές αποφασίζουν για τις μεταρρυθμίσεις και είναι υπεύθυνε για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα επωφελείται επίση και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα εξαιρετικά μέτρα υιοθετήθηκαν για την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2015 και αυτά τα έκτακτα μέτρα κατέληξαν σε πληρωμή 2,3 δισεκατομμυρίων ε, στον ειδικού σκοπού λογαριασμό για έργα και στι δύο προγραμματικέ περιόδου σημαντική επιπλέον ρευστότητα λοιπόν που δόθηκε στην ε, Ελλάδα. Για να διασφαλίσουμε την βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της για να διασφαλίσει ότι όλες οι δράσεις διοικητικές και νομικές πρέπει να ληφθούν για να ολοκληρωθούν τα έργα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, να ολοκληρωθούν ε, οι ερεσιμότητες για την περίοδο 2014-2020 και να απλουστευτεί η διαχείριση των διευθυντικών ταμείων. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα έργα ε, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα ολοκληρωθούν εγκαίρως με τα ε, εθνικά χρήματα με προθεσμία Μάρτιο του 2017 και όλες οι ε, εκ θα έχουν ε, υλοποιηθεί μέχρι τη ρυθμιστική προθεσμία που είναι τέλος του 2016. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι προσπάθειές μας για να προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ελλάδα είναι σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μια ομάδα 30 ατόμων και βοηθά επίσης την, τις ελληνικές αρχές στο να εντοπίσουν και να προετοιμάσουν τα προγράμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και μέσα στους ε, προσεχείς μήνες ε, η Ελλάδα θα αρχίσει την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Και ο Πιέχ τώρα θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη των ελληνικών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Βάλτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχα ζητήσει να με ακούσει η ομάδα εργασίας ήδη από την ημέρα που δημιουργήθηκε και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερως διότι αυτή η συνάντηση έγινε γρήγορα και πρέπει ε, και φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση εντάσσεται στις προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Ο Βάλτης παρουσίασε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βοήθεια. Και γι' αυτό εγώ ήθελα να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου στις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό πρόγραμμα. Την τελευταία φορά σας είχα παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Ήδη έχουν γίνει πολλά πράγματα. Η ανακεφαλοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έλαβε χώρα πριν τα τέλη του 2015. Σημαντικές πρόοδοι έχουν γίνει για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού, του ασφαλιστικού, για τη σύσταση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και για την ανεξαρτοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Σαφώς παραμένουν κάποια σημαντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Δεν θα πρέπει όμως να εξετάζουμε το θέμα αυτό υπό την βραχυπρόθεσμη προοπτική μόνο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματο, γιατί αυτό θα έπλητε τις δυνατότητες ανάπτυξης και θα ήταν αντιπαραγωγικό για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Τώρα, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί, όπως γνωρίζετε, να ακολουθήσουν ένα, μια δημοσιονομική διαδρομή με πλεονεσ, πλεονάσματα μισό τα 100, 1,3 και 3,5% σε σχέση με το ΑΕΠ για το 2016, 2017 και 2018 αντιστοίχως. Και ε, θα συνεχίσουν να εργάζονται, έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο ε, της συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε τον περασμένο Αύγουστο. Πολλές πρωτοβουλίες προβλέπονται σε, υπό αυτή την ε, οπτική. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο ε, νόμο σχέδιο για τα φορολογικά το 2016 και άλλα νομοθετήματα θα πρέπει να οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις. Για παράδειγμα, η συνολική μεταρρύθμιση του ε, συστήματος των συντάξεων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση του ύψους 1% του ΑΕΠ και θα, θα έρθει ως αντιστάθμισμα στο κόστος των δικαστικών αποφάσεων για ορισμένες πτυχές των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων μεταρρυθμίσεων των συντάξεων του συνταξιδοτικού. Σημαντική μεταρρύθμιση επίση ε, του ε, φόρου επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Αυτό θα φέρει έσοδα, ε, εξοικονόμηση μάλλον 1% του ΑΕΠ, μέσα από μέτρα για τη διεύρυνση τη φορολογική βάση και την μείωση των δυνατοτήτων φόρο αποφυγή. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα που αξιολογούνται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για να γίνουν και άλλε εξοικονομήσει που θα ανέρχονται σε ένα άλλο 1% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεωρούν ότι αυτή η δέσμη μέτρων του ύψου 3% του ΑΕΠ έχει ε, πολλέ πιθανότητε, ισχυρέ πιθανότητε ε, να ε, επιτρέψει την επίτευξη των στόχων του 3,5% πλεονάσματος το 2018. Το να ζητούμε επιπρόσθετες προσπάθειες από την Ελλάδα σε αυτή τη φάση των συζητήσεων είναι κάτι που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και θα απαιτούσε άλλωστε να μειωθεί ακόμα περιττέρω το βάρο του χρέου. Είδατε στα μέσα επικοινωνία μια στοιχεία και νέα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντοτε προσπαθούμε να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με αυτό τον θεσμό. Ε, συμβαίνει όμως να έχουμε ε, διαφορετικές υποθέσεις εκκίνησης, σημεία εκκίνησης και αυτό μας οδηγεί σε διαφορετικές ε, λογικές ως προς τα συμπεράσματα. πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή εκτιλήσονται στην Αθήνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το νέο Ταμείο Διωτικοποίησεων και τις Επενδύσεις ή με το άνοιγμα των αγορών ενέργειας. Να σας πω για το χρονοδιάγραμμα ότι οι επικεφαλής των αποστολών πήγαν στην Αθήνα στις 2 Απριλίου για να επιτύχουν συμφωνία γρήγορη σε τεχνικό επίπεδο, ιδανικά ε, πριν την έναρξη της Αρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή πριν το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ε, με αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, θα μπορέσουμε ίσως να έχουμε μια έγκριση στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup την επόμενη εβδομάδα και δύο-τρει εβδομάδε στη συνέχεια για τη σύνταξη των ε, νομοθετικών κειμένων και για τη διαδικασία κοινοβουλευτική έγκριση. Και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκλήρωση τη αξιολόγηση στι αρχέ του Μαΐου. Η, όπως σας είπα, η επικεφαλής των αποστολών στις 2 ε, Απριλίου θα, ε, ήρθα, ήρθα μάλλον στην Αθήνα θα συνέχισαν καθ' τη διάρκεια του περασμένου ε, κυριακού και συνεχίζουν και αυτή τη στιγμή γιατί έχει παραταθεί κατά 24 ώρες η παρουσία των επικεφαλής των διαφόρων αποστολών. Ιδανικά λοιπόν θα έχουμε ε, άτυπη έγκριση στη συνεδρίαση του Eurogroup την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε, επαναλαμβάνω, ε, δύο-τρεις εβδομάδες ε, για ε, την, τα νομοθετικά κείμενα και την κοινοβουλευτική έγκριση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκλήρωση της διαδικασίας γύρω από το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι διαχειρίσιμη αυτή τη στιγμή, όμως δεν θα πρέπει να ξαναβρεθούμε σε αδιέξοδο και γι' αυτό πιστεύουμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω την αναπόφευκτη σύγκληση μεταξύ της αξιολόγησης του προγράμματος και των διαπραγματεύσεων για το χρέος. Ε, θα ξεκινήσουμε τις τεχνικές συζητήσεις ήδη στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες και ε, σε σχετικό υπουργικό επίπεδο. Έχουμε διάφορες επιλογές μπροστά μας και η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι να διευκολύνει τις συζητήσεις όσο περισσότερο ε, μπορεί. Αυτά προς το παρόν και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και οι δύο παρουσιάσεις επικυρώνουν το ενδεχόμενο συμφωνίας και την αναγκαιότητα της συμφωνίας. Είναι πολύ θετική αυτή η επικύρωση ότι και η επιβεβαίωση, η διαβεβαίωση ότι και η Κομισιόν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα συμφωνούν ε, στο προσδιορισμό του δημοσιονομικού στόχου, ο οποίος είναι και αποδεκτός από τις ελληνικές αρχές. Οπότε δύσκολα θα μπορέσουν να τον αμφισβητήσουν άλλα θεσμικά όργανα. Ξεκινάμε από τις ερωτήσεις. Ο κύριος Κέτσος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η διαφορά σας ε, στις απόψεις είναι στατιστικής ή πολιτικής φύσης. Αφορούν πολιτικές δηλαδή που πρέπει να ακολουθηθούν, διότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει με δραματική εικόνα αυτές τις διαφορές η ελληνική κυβέρνηση έχει αναφερθεί σε επιθετική πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας μάλιστα ισχυρίζεται ότι εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα μια χαρά χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας αναλύσετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε, να καλύψετε αυτές τις διαφορές γιατί είναι ε, ύψη της σημασίας. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο δηλαδή τα χρήματα που πρέπει να καταβάλει το κράτος ε, στους πιστωτές, αλλά και ε, το πώς θα λειτουργήσει η ιδιωτική ε, οικονομία. Όταν λεξιπρόθεσμα αυξάνονται ε, όταν συζητάμε λοιπόν για μια συμφωνία μέσα στι επόμενε λίγε εβδομάδε, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση τη ελληνική οικονομία, θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο ακριβεί. Ευχαριστώ. Ποιο θα ήθελε να ξεκινήσει. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Πράγματι, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συνεργαστεί στενά. Το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αποτελεί αναπόσπαστο ε, μέτοχο, ε, κομμάτι της πρώτης ε, ανα, αναθεώρησης, της πρώτης αξιολόγησης ε, όσον αφορά τους στόχους και τα μέτρα που απαιτούνται για την επιτεύξη των στόχων του προγράμματος. φυσικά επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων όσον αφορά ε, τις ε, εκτιμήσεις, τι προσπάθειες ακριβώς θα χρειαστούν για την επιτευξή των δημοσιονομικών στόχων. Υπάρχουν κάποιες διαφορές επί λεπτομεριών για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα μπορούν να γεφυρωθούν. Υπάρχουν και κάποιες ε, τυπικές διαφορές. Εμείς προετοιμάζουμε το δικό μας το μνημόνιο, το δικό μας έγγραφο, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκπονεί ένα άλλο έγγραφο δικό του, βάσει των δικών του διαδικασιών. Αλλά το ίδιο είχε συμβεί και σε παλαιότερα ελληνικά προγράμματα, όπως και σε προγράμματα με άλλες χώρες. Διότι για νομικούς λόγους το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ε, αναφέρεται σε άλλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εμείς ας πούμε αναφερόμαστε στην, ε, είμαστε υπολόγοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λοιπούς, οπότε οι διαδικασίες που ακολουθούμε είναι διαφορετικές. Αλλά θα έλεγα ότι συνεργαζόμαστε πολύ επικοδομητικά και κάποιες διαφορές ε, εκτίμησης ε, πιστεύουμε ότι μπορούν να γεφυρωθούν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, Σίγουρα μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα έχουμε την επόμενη εκταμίευση ε, στο πλαίσιο του προγράμματος. Έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα. Η εκταμίευση ακολουθεί την αξιολόγηση. Αυτός και ακριβώς είναι και ο σκοπός και δεν αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν ο Πιέρ θα ήθελε να, λύσει κάτι, να πει κάτι άλλο. Ναι, ε, συμφωνώ απολύτως με τον Βάλτης και για τα δύο αυτά θέματα. Δεν υπάρχει διαφορά στην πολιτική προσέγγιση και δεν υπάρχει θέμα τακτικής. Δεν υιοθετούνται τακτικές όταν πρόκειται για ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχουν θεσμικές διαφορές, διαφορές επί της διαδικασίας, στατιστικές διαφορές οι οποίες ε, βρίσκονται υπό την ε, διαιτησία, αν θέλετε, των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω η βούληση όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όλων των θεσμών γενικότερα είναι να συνεχίσουν να εργάζονται ε, μαζί γιατί είναι το καλύτερο και για τα κρατη και για την Ελλάδα. Δεν θέλω λοιπόν να υποκύψω σε αυτές τις ε, ε, διάφορες εικασίες που προβάλλουν τα διαφορετικά μέσα ενημέρωσης για να δείξουν τάχα διαφορετικά μνημόνια. Υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, υπάρχει μία συμφωνία, οι θεσμοί είναι δίπλα-δίπλα παρόλο που οι παράμετροι ενδεχομένως είναι διαφορετικές ε, σε επίπεδο στατιστικών δεδομένων και άλλων. Δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα για την ελληνική οικονομία σήμερα και άπαξ και ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση θα είμαστε σε θέση να προβούμε στην εκταμίευση την προβλεπόμενη ε, βάση του προγράμματος. Όμως οφείλουμε επίσης να παρακολουθούμε στενά την, την ε, κατάσταση της ρευστότητας, γιατί δεν θα είναι επαόριστον η ανυπαρξία προβλήματος ε, ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό. Υπογραμμίζω την έκφραση το συντομότερο δυνατό. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε. Και Ε, αν χρειάζεται χρόνος για να το ολοκληρώσουμε, να δώσουμε αυτό το χρόνο. Εάν δεν χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί, τότε να μην ε, προχωρήσει ενδεχομένως χωρίς λόγο. Ευχαριστώ. Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Επίτροπη. Μιλάμε για μια οικονομία που έχασε 40% του δυναμικού της τα τελευταία χρόνια και τώρα βρίσκεται σε στασιμότητα. Μιλάμε για ένα κράτος μέλος που προφανώς σύμφωνα με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να υλοποιήσει τα προγράμματα μεταρρύθμισης και μιλάμε για μια χώρα που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην πολιτική μας στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο θέμα του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το ζήτημα ε, του μεταναστευτικού. Η Ευρώπη είναι γεμάτη απειλές ε, θα αναφέρω απλώ την 23η Ιουνίου και την απόφαση που πρέπει να ληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Δεδομένη τη σοβαρότητα τη κατάσταση, μπορείτε να εγγυηθείτε και να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι θεσμικό. Όταν στη συνάντησή μας στην Αθήνα συναντήσαμε είτε την τράπεζα, είτε το ΤΑΙΠΕΔ, είτε ε, ε, ιδιώτες εμπλεκόμενους, όλοι τόνισαν ότι είναι σημαντική αυτή η χρονική στιγμή και πρέπει να τονώσουμε την οικονομία, να προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν είναι σίγουρα, αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε, ότι το Eurogroup εκφράζεται με μία φωνή και ποιο είναι το εμπόδιο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο να είναι στην ίδια, στο ίδιο πλοίο μαζί μας ώστε να μπορούμε να βρούμε κοινέ λύσεις. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε για λύσεις από εδώ και πέρα. Well, uh, as, uh, Λοιπόν, ε, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, πράγματι η Ελλάδα έχει περάσει μακροχρόνια και βαθιά ύφεση. Και πράγματι τα πράγματα είχαν αρχίσει να βελτιώνονται το 2014, όπου είχε επιστρέψει η ελληνική οικονομία στην ανάπτυξη, όπου η ανεργία είχε αρχίσει να μειώνεται, όπου η Ελλάδα κάλυπτε και ε, πετύχαινε τους δημοσιονομικούς στόχους, ε, είχε καθυσχάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αρχές του περσινού έτους περιμέναμε ανάπτυξη 2,5% για την Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε, οι πολιτικές εξέλιξεις όμως ε, την ανάγκησαν να αλλάξει δρόμο και ε, επανήλθε η οικονομική αστάθεια ε, και δυστυχώς η οικονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Ελήψη λοιπόν οικονομικής ε, σταθερότητας στο πρώτο εξάμεινο του 2015 η Ελλάδα δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην ανάπτυξη και πράγματι ε, οι χειμερινέ μα οικονομικέ οικονομικές προβλέψεις έδειχναν μηδενική ανάπτυξη στην Ελλάδα πέρυσι αλλά όπως είπαμε τα στοιχεία από την Ελλάδα δείχνουν ε, πιο θετική πορεία και ίσως το Μάιο το αποτέλεσμα που θα είναι καλύτερο. Δείχνει όμως και κάτι άλλο, ότι η ελληνική οικονομία ε, δεν έχει τις δυνατότητες, ε, ε, τις λείπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε μόλις επανέλθει η οικονομική σταθερότητα που αποτελεί βασικό ορόσημο, η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να ανακάμψει. Και εκεί, όπως είπα πριν από ένα εξάμεινο περίπου, εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε κάποιες θετικές εκπλήξεις. Πράγματι όμως, όπως είπατε και εσείς, ε, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλαπλές ε, κρίσεις. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν πλήρως την πολυπλικότητα της κατάστασης και την ανάγκη εξεύρεση μιας λύσης. Αλλά η λύση φυσικά εξαρτάται και από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ε, όπως αυτές προβλέπονται στο μνημόνιο. Όσον αφορά το Eurogroup, ρωτάτε αν μιλάει με μία φωνή, θα έλεγα ναι. Λάβαμε σαφή εντολή από το Eurogroup ήδη από τον Αύγουστο πέρυσι και από τα όσα μαθαίνουμε από τους συναδέλφους μας στο Eurogroup, στο Eurogroup είναι ότι εμένουν σε αυτή την εντολή και σε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Μοσκοβησέ. Εν συντομία, προς την ίδια κατεύθυνση και εγώ θα κινηθώ. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια ή τακτικές και τακτικισμοί σε τέτοιου είδους θέματα. Αυτό δεν είναι δυνατό. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το πλαίσιο. Η Ελλάδα χρειάζεται να επανέλθει στην ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ και μάλιστα γνωρίζουμε και το ύψος της πρόκλησης την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα με την κρίση των προσφύγων, με το προσφυγικό. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις δεν μπορούν να είναι πολιτικές, δηλαδή υποκειμενικές. Ε, δουλεύουμε πάνω στη βάση ενός Memorandum of Understanding, ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο αποτελεί και τον οδικό μας χάρτη. Είναι πολύ σημαντικές οι πρόοδοι που έχουν καταγραφεί στη διαπραγμάτευση και φαίνεται ότι υπάρχει κοινή εκτίμηση από πλευρά θεσμών και δεν είμαστε ακόμα στο καταληκτικό σημείο, εξού και υπάρχει ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ε, πάνω σε αυτή την ε, ε, σε αυτά τα αντικειμενικά σημεία. Επίσης δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, η κατάσταση μπορεί να γίνει ανησυχητική και όσο συντομότερα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις τόσο γρηγορότερα θα έρθει η εκταμίευση και τόσο γρηγορότερα θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και θα μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά δεν παίζουμε με αυτά και γι' αυτό λέμε ας ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό, δηλαδή γρήγορα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι εφικτό, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειε. και ε, λέω ότι ιδανικά, ε, αναλόγω με τι εξελίξει, μπορούμε στα τέλη αυτή τη εβδομάδα ή και στην επόμενη εβδομάδα να ολοκληρωθούν κληρωθούν οι διαδικασίες για να πάμε μετά στο Eurogroup και να ακολουθηθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μοσκοβισή. Διέρεσε, διέρευσαν τα πρακτικά μια συζήτηση του διεθνού Νομισματικού Ταμείου και το περιεχόμενο δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικό για την Ευρωζώνη. Αναφέρεται σε αυτά τα πρακτικά ότι η Ευρωζώνη ε, θα ε, θα έκανε παραχώρηση ε, για την Ελλάδα, δηλαδή ότι η Ευρωζώνη δεν έχει κάποια κόκκινη γραμμή όσον αφορά τις απαιτήσει προς την Ελλάδα. Η ερώτησή μου είναι απλούστατη. Έχετε κάποια κόκκινη γραμμή και ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή σας. Και πάλι θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω γιατί να σας μιλήσω για τέτοιου είδους έγγραφα και διαρροές είναι πράγματα τα οποία ε, δεν σχολιάζω και δεν εξετάζω. Μπορώ να σας πω ότι είναι κοινή η δουλειά και η εξέταση από τους θεσμούς είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχουν ούτε κόκκινες, ούτε κίτρινες, ούτε άσπρες, ούτε μπλε γραμμές. Υπάρχει κάτι πολύ απλό. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ο οποίος είναι κοινό για όλους, το μνημόνιο κατανόησης. Και αυτός ο οδικός χάρτης δεν επιδέχεται υπερβολικά υποκειμενικών ερμηνειών. Πιστεύω. Δεν θα πρέπει κανείς να έχει υπερβολικά πολιτική προσέγγιση με την κακή έννοια του όρου ή υπερβολικά πολεμική προσέγγιση με την καταστροφική έννοια του όρου. Μιλούμε για μια χώρα η οποία έχει χάσει το 30% του ΕΠΤΗ σε κάποια χρόνια. Πρέπει να κάνει προσπάθειες, αλλά χρειάζεται απεγνωσμένα την ανάπτυξη. Πρέπει να κάνουμε όλοι προσπάθειες. Και ας μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι ρόλων του ποιο είναι σοβαρός και ποιο δεν είναι. Οι θεσμοί θα φτάσουν στα τέλη, στο τέλος της διαδρομής μαζί, έχουν διανύσει αυτή την απόσταση μαζί. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι που θα πρέπει να συγκλίνουν γύρω από την ίδια πραγματικότητα βάσει των ίδιων κανόνων και ε, βάσει του ιδίου κειμένου που είναι το μνημόνιο κατανόησης ε, που ε, συντάχθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ο ο Υπουργό Σόιμπλε έχει δηλώσει ότι είναι πεπισμένο ότι μπορεί να βρεθεί λύση και συμφωνώ απολύτω μαζί του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και όλοι πιστεύουμε ότι θα βρεθεί μια ε, λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάχ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων, ξέρετε. Έχω μία ερώτηση στο πλαίσιο που δημιουργεί προβλήματα η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ορισμένες χώρες. Έχετε την αίσθηση ότι ε, τηρείται αυτή η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, γιατί εμείς από τα κράτη-μέλη επιθυμούμε την ε, άψογη εφαρμογή του περιεχομένου της συνθήκη. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε, γιατί για μένα η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο αέρας που αναπνέω σχεδόν, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι σας ανησυχεί. Ουσιαστικά δύο είναι οι ερωτήσει μου. Η μία μετά από τη δημιουργία τη Τρόικα, ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε σχέση με του υπόλοιπου και συχνά λέει ο κ. Ντράγκη μπροστά μα ότι θεωρεί ότι η Κεντρική Τράπεζα ε, προσφέρει αρρωγή στα άλλα θεσμικά όργανα, θεωρείται ότι έτσι λειτουργεί. Και πέραν ε, αυτού δεν νομίζετε ότι είναι πολύ σημαντικό δεδομένο των σημερινών συνθήκων. Αν λέτε ότι είναι ο αέρας που αναπνέεται θα διαβάζετε και εφημερίδες όπου θα διαβάζετε τα ίδια όπως και εγώ. Η ερώτησή μου είναι πολύ σοβαρή. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαμε μια διαρκή αντίδραση ε, για τα διάφορα μακροπρόθεσμα σχέδια. Ε, υπάρχουν κάποιε αντιδράσει όπου διάφορε κυβερνήσει ε, προσπαθούν να επηρεάσουν όλο και περισσότερο την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πάρω τι ερωτήσει σα ε, ανάποδα, αν κατάλαβα καλά, να σα δώσω κάποιε διευκρινήσει. Όταν λέω ότι είναι ο αέρα που αναπνέω, πιστεύω πράγματι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβάλλει ουσιαστικά στο μέλλον της Ευρωζώνης και τρέφω τεράστιο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο τα λόγια και οι πράξεις του Μαρίο Ντράγκη βοήθησαν να απαγιωθεί ε, η Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι κανένας, ούτε καν όσοι επέμειναν παλιότερα για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χρειάζεται να ανησυχούν. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαδικασίες ε, ε, που τηρούνται από όλους και πρέπει να τηρούνται από όλους όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνει η ίδια. Έτσι λοιπόν ε, δεν μπορούμε να ανεχθούμε καμία αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερη ερώτηση τώρα, ως, αν δούμε ε, τις λεπτομέρειες λειτουργίας των θεσμών της Τρόικας, ανέκαθεν υπήρξε σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάπως, έναν κάπως ιδιαίτερο ρόλο και υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος συνομιλητής. Ωστόσο δεν πιστεύω ότι ακολουθούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρώ ότι ήταν συντονισμένες οι ενέργειες αρκετά καλά. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σε δεύτερη μοίρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι είχε δευτερεύοντα ρόλο. Αλλά ναι, η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή ανέλαβε τις ευθύνες της όπως ε, οδηγός ε, της όλης διαπραγμάτευσης. αλλά ε, σεβόμενοι όλους τους υπόλοιπους ε, το Διεθνές το Δανείο λειτουργεί κάπως διαφορετικά όλα αυτά συντονίστηκαν μεταξύ τους και έτσι λειτουργήσε το, η όλη διαδικασία ε, well, yes, just... Ο κύριος Ντομπρόφσκης συμπληρώσω και εγώ αυτά που μόλις είπε ο Επίτροπος Μοσκοβισή και βέβαια σεβόμαστε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα, ε, και θα πρέπει να τηρούνται από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με στενή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπου αυτό είναι εφικτό. Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε σύμφωνα με τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα, που προβλέπει και τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και όντω ήταν πολύ σημαντικό ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υποστήριξε ε, το τομέα των τραπεζών, την ρευστότητα κλπ. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προ τον κύριο Μοσκοβισή. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ απολύτω μαζί σα ότι δεν υπάρχει καιρό για χάσιμο από τη στιγμή που, όπω και εσεί σημειώνετε, έχει επιτευχθεί μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας αλλά και στις συζητήσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα σημεία που απομένουν να γεφυρωθούν για την ολοκλήρωση αυτής της περίφημης πρώτης αξιολόγησης. Από την πληροφόρηση που εγώ έχω, η ελληνική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει μία πρόταση για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος με τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ταμείου. Αμφιβάλλω αν στις χώρες σας θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μια τέτοια μεταρρύθμιση, η οποία εξασφαλίζει την εξοικονόμηση τη συμφωνημένη του 1% του ΑΕΠ με την εξής αναλογία. 75% αυτών των περικοπών αυτής της οικονομίας από περικοπές συντάξεων κατάργηση των πρόορων συνταξιοδοτήσεων και περικοπές στις συντάξεις τις επικουρικές, supplementary pensions, και το άλλο 25% από μια μικρή προσωρινή αύξηση των εισφορών των κοινωνικών εργοδοτών και εργαζομένων, στην οποία σημειώνω ότι υπάρχει κοινωνική συνένεση, καθώς έχουν συμφωνήσει και όλες οι οργανώσεις των Ελλήνων εργοδοτών γιατί διαφωνείτε με αυτή την πρόταση που εξασφαλίζει την υλοποίηση της συμφωνίας με την συμμετοχή και στο μείγμα αυτό και μιας μικρής προσωρινής άξης εισφορών που δέχονται οι Έλληνες εργοδότες. Το δεύτερο, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει μια πρόταση που λέει να εξαιρεθεί για ένα μικρό εύλογο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, η προστασία μόνο των δανείων που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία. Δηλαδή ένας μικρός επιχειρηματίας που δανείστηκε για να σώσει την επιχείρησή του και έβαλε ως ενέχειρο την πρώτη κατοικία, να μην την χάσει αλλά να έχει μια προστασία μικρή για ένα, ενάμιση χρόνο. Διαφωνεί η Κομισιόν σε αυτό. Διότι αν αυτά είναι οι διαφορές, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται μια προσπάθεια να συναντηθείτε στα μισά της γέφυρας. Δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες ε, της συζήτησης γιατί είναι διαπραγματεύσεις που εκτιλήσονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα την ώρα που μιλάμε. Βεβαίως είμαι σε επικοινωνία με τους επικεφαλεί των αποστολών μας και ε, μιλώ, συνομιλώ επανειλημμένως πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον Υπουργό ε, κύριο Τσακαλώτο. Την τελευταία φορά που του μίλησε ήταν Σάββατο βράδυ σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών. Να σα πω ότι ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές προόδοι για το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού, του ασφαλιστικού, για την ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και Είμαστε σε συζητήσεις για την ανεξάρτητη αρχή, αν θέλετε, εσόδων δηλαδή και είμαστε σε συζητήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η αίσθηση που έχουμε, που έχουμε αποκομίσει είναι ότι σήμερα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα μας επέτρεπε να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει. Θα συνεχιστούν οι συζητήσει, θα έχουμε αποτελέσματα απόψε και στη συνέχεια θα έχουμε τι επόμενε μέρε χρήσιμε ανταλλαγέ απόψεων πριν πάμε στην Ουάσιγκτον. Αλλά και στην Ουάσιγκτον, στην Νεαρήνη Σύνοδο, θα έχουμε ε, χρήσιμε ανταλλαγέ απόψεων. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε μία ε, γραμμή που μας καθοδηγεί όλοι που είναι η τήρηση του μνημονίου κατανόησης των απαιτήσεων σε σχέση με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα ε, που ε, πρέπει κανείς να ε, φέρει. Τώρα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να σας πω ότι βελτιώνεται το πλαίσιο. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ζητήθηκε από τις τράπεζες να, πάρουν, να κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τράπεζες έχουν συγκεκριμένα σχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και για την πώληση αυτών σε εταιρείε. Όμως το νομικό πλαίσιο στηρίζει όλο και περισσότερες, περισσότερο αυτές τις δράσεις. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συγκεκριμένες ε, δράσεις σχεδιάσει. Έχει αλλάξει ο κώδικας πολιτικής δικαιονομίας. Έχει αλλα... Ε, είναι κάπως απαξιωμένη η ελληνική νομοθεσία για την κήρυξη χρεοκοπίας των επιχειρήσεων. Παραμένει η δουλειά που πρέπει να γίνει για να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν τα νούμερα των τραπεζών σε σχέση ε, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πρέπει να έχουμε επιχειρησιακούς στόχους για τις τράπεζες έτσι ώστε να μειωθεί το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε κάθε συστημική ε, τράπεζα. Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας που ε, έχει ψηφιστεί, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2016 λόγω της αποχής των δικηγόρων είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί όλη η νομοθεσία και να εφαρμοστεί στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και για το προηγούμενο ερώτημα βέβαια, δηλαδή πολύ καλή πρόοδος και σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά όχι ο πλήρης πρόοδος ολοκληρωμένη. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και οι επίτροποι που ήρθατε σήμερα στη συνεδριασή μας. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον θέλω να επανέλθω σε αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος. Στη συζήτηση για τη σταθεροποίηση του συνταξιοδοτικού προτείνει η ελληνική κυβέρνηση ε, τρία χρόνια με 1,5% των εισφορών και ε, οι θεσμοί και η Επιτροπή δεν συμφωνούν. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ε, ποιος είναι ο λόγος που δεν συμφωνούν. Επίσης, η Επιτροπή μα έχει πει σε προηγούμενε συνεδριάσει στην Επιτροπή μα ότι οι θεσμοί δεν ε, θα ζητήσουν να θυγεί το ονομαστικό επίπεδο των συντάξεων. Τώρα ζητάτε μείωση ονομαστικά των συντάξεων και για το Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων στην Αθήνα ο κύριος Σταθάκης μας είπε ότι ο στόχος των 50 δισεκατομμυρίων δεν ήταν ρεαλιστικός. Είπε ότι για φέτος ο στόχος θα είναι 2,5 δις και το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να φτάσει 6,5 ε, δις ως στόχο. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Εσείς ως Επιτροπή συμφωνείτε με το στόχο των 50 δις που αναφέρεται στο μνημόνιο ή συμφωνείτε με τα στοιχεία τα οποία μόλις σας ανέφερα. Uh, okay. So, uh, Λοιπόν, ο κύριος Ντομπρόφσκης, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το συνταξιοδοτικό. Όπως ήδη είπε ο Πιέχ, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εν εξελίξη. Η ελληνική κυβέρνηση όντως υπέβαλε μια συνεκτική πρόταση πριν από κάποιους μήνες και συμπεριλάμβανε και προσωρινές αυξήσεις στις συνταξιοδοτικές εισφορές. Αυτά είναι σημεία τα οποία βρίσκονται στη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί και στο μνημόνιο για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος για να απλουστευτεί το σύστημα αυτό και για να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένο να είναι οι συντάξεις περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τις εισφορές ε, των ε, εργαζομένων κατά τη διάρκεια ε, της ζωής τους. Αλλά όπως σας είπα οι συζητήσεις βρίσκονται εν εξέλιξη και δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τώρα για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Όντως όσον αφορά τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσει, αναμένουμε έσοδα 2 2,5 δις ευρώ φέτος. που θα πρέπει να το συγκρίνουμε με τα 250.000 ευρώ πέρυσι και μέχρι το 2018 ο συνολικός στόχος είναι 6,2 δις για τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων. Φιλόδοξος αλλά εφικτός ο στόχος εάν η κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει την αποφασιστικότητα που έδειχνε τους τελευταίους μήνες. Ο στόχος των 50 δις που αναφέρεται είναι περισσότερο μακροπρόθεσμος στόχος. Η θέση της Επιτροπής υπάρχει στο μνημόνιο, όπως συμφωνήθηκε τον Αύγουστο. Και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων σαφώς αποτελεί τμήμα της όλης συμφωνίας. Δημιουργήθηκε ε, ως ε, τμήμα της δεύτερης ομάδας προαπαιτουμένων. Η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε το Ταμείο για να είναι ενεργό το 2016 και θα πρέπει η νομοθεσία να έχει εγκριθεί ως τμήμα των συζητήσεων της πρώτης αξιολόγησης και να λυθούν τα μέτρα υλοποίησης. Δηλαδή, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή εκ παραλλήλου σε πολλά πεδία. Σχέδιο νομοθεσίας για το Ταμείο, οικονομικό μοντέλο και απαιτήσει ε, κεφαλαίου. Ποιε ε, επιχειρήσεις θα μεταφερθούν στο Ταμείο, πολιτική λειτουργία του Ταμείου, επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Συνεχίζεται λοιπόν η εργασία σε όλα αυτά τα πεδία εκ παραλίλου και νομίζω ότι ε, βρισκόμαστε σε καλή πορεία όσον αφορά το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Δεν ξέρω ποια θέλει να πει κάτι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Κύριε Άνεμαντς. κύριος Θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο το ερώτημα του κυρίου Λούκας. Ε, ε, ας απαντήσει ο κ. Μοσκοβισή, αλλά θα την κάνω την ερώτηση στα Ολλανδικά. Η συζήτηση ε, που προέκυψε από το Wikileaks ε, για τους διευθυντές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την αφήσατε στο πλάι, την κρύψατε, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα όταν μιλάμε για το ελληνικό χρέος. Εδώ θα σας διαβάσω το εξής που υπόθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι συμφωνούν ε, για ένα πράγμα και μετά το ξεχνούν την επόμενη μέρα. Έχουμε πει επανειλημμένω ότι δεν κάνουν αυτά ε, που λέμε, δεν λειτουργεί. Τίποτα δεν τους αρέσει, όλα μπορεί να αλλάξουν ε, εφόσον το θέλουν οι αρχές. Σας διαβάσα αυτό το απόσπασμα και έχω ξανακάνει την ερώτηση σε έναν διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μου λέει ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφόσον συναυθεί η συμφωνία με την Ελλάδα. Οπότε το ερώτημα είναι τι άποψη έχει το, Ευρωπαϊκ... το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φαίνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα δίνει τη συμφωνία της, αλλά τι θα γίνει το ζήτημα πρέπει να επιληθεί από πλευρά κομισιών, αλλά είναι πολιτικό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν αφού βρίσκονται εδώ σήμερα οι Επίτροποι ε, συμφωνείτε με αυτή την αναγνώριση της ε, διαγραφής του ελληνικού δανείου σε περίπτωση συμφωνίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μην σχολιάσω, επαναλαμβάνω, αυτή τη διαρροή γιατί δεν γνωρίζω την πρόλευσή της, ε, την πρόλευσή της και δεν ε, μπορώ να γνωρίζω έτσι την αξιοπιστία της. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι εμείς ε, ε, αποσκοπούμε σε συμφωνία, συμφωνία καθολική. Και φυσικά, δεδομένου αυτού, έχουμε συνείδηση του γεγονότος ότι θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια σύνδεση μεταξύ της μείωσης της εξυπηρέτησης του ελληνικού δανείου και του ίδιου του προγράμματος. Ε, έχει υποθεί, αναφέρεται στη συμφωνία του Νοεμβρίου 2012 του Eurogroup υπό συγκεκριμένου όρου. Ποια στιγμή θα αρχίσουμε να μιλάμε για το χρέος, ε, έρχεται αυτή τη στιγμή αναμφίβολα. Ε, και η Κομισιόν διατίθεται να πράξει κάτι τέτοιο, έχοντας γνώση του γεγονότος ότι ελέγξτε όρεξη έχουν τα κράτη-μέλη, για να μην το πω περισσότερο, για haircuts, για περικοπές, για κούρεμα το ζήτημα της υλοποίησης είναι πολύ σημαντικό. Ε, ξέρετε, το να υιοθετήσουμε μια συμφωνία είναι ένα πράγμα, το να την υλοποιήσουμε είναι κάτι άλλο. Ε, η λέξη implementation είναι η λέξη κλειδί για μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι αν δεν υλοποιηθεί επαρκώς η συμφωνία, γιατί ούτως ή άλλως γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια συμφωνία. Ε, για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Αυτό συμφέρει και την Ελλάδα. Ε, διαφορετικά εμείς δεν θα είχαμε ξεκινήσει τέτοια διαδικασία, ούτε θα είχαμε δεσμευτεί. Επίσης να επαναλάβω, ας μην προσπαθήσουμε να ασκήσουμε υπερβολική να τραβήξουμε στα άκρα τα σενάρια και το τι ρόλο παίζει το καθεθεσμικό όργανο. Οι σχέσεις μας είναι απλές. Έχουμε ένα κοινό οδικό χάρτη, το μνημόνιο, έχουμε απόψεις θεσμικές ως αφετηρίες ε, ίσως διαφορετικές ε, ίσως ο τρόπος που βλέπουμε τα στατιστικά μοντέλα να μην είναι ακριβώς ο ίδιος, αλλά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τους θεσμούς, διότι όλοι μαζί εργαζόμαστε σε τελική ανάλυση και όλοι μαζί θα συνάψουμε αυτή τη συμφωνία. Οπότε έχουμε πολύ συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης ε, του θέματος όλοι μαζί. Thank you. Now we Ευχαριστούμε. Τώρα το, η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Βαμβαϊτσέκερ. Καταλαβαίνω απολύτως και νομίζω ότι είναι συνετό το ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε τις διαρροές. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα ερωτηματικά. Είπατε ότι τελικά θα υπάρξει κάποιος συμβιβασμός, όντως. Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι θα έχουμε ένα συμβιβασμό που θα βασίζεται σε ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις, σε υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα και σε μια υπερβολικά φιλόδοξη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και νομίζω ότι μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης αυτός ο διανοητικά νοθρός συμβιβασμός είναι παγίδα και ο ρόλος του Δουνουτού είναι να μας βοηθήσει να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή. Διερωτώ με πώς μπορείτε να δείξετε στους ψηφοφόρους μας ότι δεν θα είναι νοθρός διανοητικά συμβιβασμός αυτός στον οποίο θα καταλήξετε το καλοκαίρι, αλλά θα βασίζεται σε ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες χρειάζεται η Ελλάδα και μια ρεαλιστική αξιολόγηση για το τι είναι πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα και ρεαλιστική ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ο κ. Ντομπρόφσκης για την ερώτησή σα, θέλω να απαντήσω ότι όντω εργαζόμαστε επικοδομητικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στις εκτιμήσεις, οι οποίε όμως μπορούν να γεφυρωθούν και νομίζω ότι αυτό και θα καταφέρουμε να κάνουμε. Τώρα, για το θέμα του ε, υπερβολικού πρωτογενούς πλεονάσματος. Το πρωτογενές πλεονάσμα υπάρχει στο μνημόνιο του περασμένου Αυγούστου και πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2018. 3,5% του ΑΕΠ πρέπει να επιτευχθεί ως πρωτογενές πλεόνασμα, ε, δηλαδή 1,5% του ΑΕΠ λιγότερο από το προηγούμενο ελληνικό πρόγραμμα, το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα, που προέβλεπε ως μεσοπρόθεσμο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε στις διαπραγματεύσεις και αυτό ανακολουθεί η Επιτροπή με βάση την εντολή που μας έχει δώσει το Eurogroup. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, είπατε ότι είναι ανεπαρκείς οι μεταρρυθμίσεις. Οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις για την ελληνική οικονομία είναι βεβαίως απαραίτητες ε, και εργαζόμαστε εντατικά με τις ελληνικές αρχές προς την κατεύθυνση αυτή. Σημειώστε παρακαλώ ότι ήταν εμπροστοβαρές το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων συμφωνήθηκαν ε, και ε, θεσπίστηκαν σε νομοθεσία αρκετές μεταρρυθμίσεις ε, και άρχισαν να υλοποιούνται πριν από την εκταμείευση χρημάτων προς την Ελλάδα και ελήφθησαν και περαιτέρω σημαντικά μέτρα στο πλαίσιο της πρώτης και της δεύτερης δέσμης προαπαιτούμενων μέτρων. Δηλαδή, η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσει για τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τώρα, αλλά βεβαίω και πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα και χρειάζεται και καθοδήγηση για το τι πρέπει να επιτευχθεί. Όσον αφορά την ανάλυση βιωσιμότητα του χρέους, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ρεαλιστική ανάλυση βιωσιμότητα, όπως είπατε και όχι πολύ φιλόδοξη και η ανάλυση ε, την οποία κάναμε πέρυσι τον Αύγουστο έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δεν θα την αποκαλούσα φιλόδοξη, ε, αισιόδοξη αυτή την ε, ανάλυση διότι οι οικονομικές προοπτικές από πέρυσι και η οικονομική πρόοδος ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους πέρυσι τον Αύγουστο. Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική και δεν είναι υπερβολικά απεσιόδοξη για το μέλλον και η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους συνδέεται άμεσα με τα μέτρα που αφορούν το χρέος και είναι περιορισμένο το περιθώριο ελιγμών όπως ήδη είπε ο Πιέχ. Το Eurogroup ήδη έχει συμφωνήσει να επανέλθει σε αυτό το θέμα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ε, χωρίς να μιλάμε για ονομαστική, ονομαστικό κουρέμα του χρέους. Δύο λόγια για αυτά που είπε ο Βάλτης. Θέλω πραγματικά να εξαλείψω από το προσκήνιο αυτή την ιδέα ότι υπάρχει ας πούμε ένα παιχνίδι ρόλων από πλευράς θεσμών. Η οκνηρή με, η μεν και η σοβαρή η ε, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Απορρίπτω κατηγορηματικά τέτοιου είδους εικασίες και θα φτάσουμε σε ένα τελικό σημείο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι αυτό απαραίτητο. Στηρίζω επίσης τις ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα η εκτίμησή μας είναι ότι αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διάφορες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό, στο συνταξιδωτικό και στα άλλα μέτρα, μπορούμε να έχουμε μια δέσμη μέτρων 3% του ΑΕΠ και αυτό θα επέτρεπε να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2018. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως διαφορετική για το σημείο, γιατί το σημείο κίνησης της για το 2015 είναι κάπως πιο αυστηρά, αυστηρό. Ε, δεν είναι στατική προσέγγιση. Η αίσθηση μου είναι ότι η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακριβής, είναι η σωστή. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με ρεαλιστικό ε, τρόπο. Δεν είναι το σημείο κίνηση ούτε υπερβολικά αισιόδοξο ούτε υπερβολικά απεσιόδοξο. Είναι ακριβές. Τώρα το θέμα είναι να έχουμε στατιστικά στοιχεία που μπορούν να ε, συγκεράσουν αυτές τις δύο εκδοχές με αντικειμενικό τρόπο. Εάν για παράδειγμα προέκυπτε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφάλουμε ε, ως προς τα στοιχεία, τότε θα μετατεθούν οι δύσκολε αποφάσει για πιο μετά και δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουμε νυφαλιότητα, αντικειμενικότητα και αυτό προσπαθούμε να έχουμε και να περάσουμε σαν γραμμή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη σωστή υπόθεση εργασίας και αυτό επαληθεύεται και από τους λοιπούς ε, θεσμούς. Δεν υπάρχει διαίρεση μεταξύ Ευρώπης και Δουνουτού και σήμερα όλοι ε, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λοιποί έχουν τις ίδιες εκτιμήσεις όπως εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επαναλαμβάνω δεν θα μας χωρίσει κανείς, δεν θα μας διαιρέσει είναι ένα, θα ήταν ένα τεράστιο σφάλμα το οποίο δεν θα διαπράξουμε. Thank Ευχαριστούμε και έχουμε και τα νούμερα που όπως φαίνεται είναι καλύτερα από ό,τι αναμέναμε όπως είπε ο Βάλτης ε, κύριε Πρεβόνς Μπερές ε, ευχαριστώ πολύ ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα και εγώ συμμετείχα στην αποστολή στην Αθήνα θα ήθελα να πω καταρχάς ε, στην Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται διαβεβαιώσεις. Να σας πω πόσο μεγάλη εντύπωση μας έκανε ο εκπρόσωπος επιτόπου ο κ. Κοστέλο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Είχαμε μια επικοδομητική, εποφελή ε, ανταλλαγή απόψεων γεμάτη εμπιστοσύνη. Μου φάνηκε ότι υπάρχει κοινή βούληση στην αντιπροσωπεία ε, Υπό αυτές τις συνθήκες ε, ο κύριος Μοσκοβησί απάντησε εν μέρη, είπε δεν θα μας διαχωρίσει κανείς. Αλλά σε περίπτωση συζήτησης ε, μεταξύ, όταν υπάρχει συζήτηση μεταξύ των ε, θεσμών και μετά αποστολή στην Αθήνα, όσοι έχουν νομιμοποιηθεί και έχουν δεσμευτεί επί τόπου για να ηγηθούν της όλης διαδικασίας, είναι ουσιαστικά οι θεσμοί τη Ένωση. Αυτοί έχουν λάβει την εντολή. Οπότε έτσι ξεκινάει αυτή η διαπραγμάτευση όπου προφανώς το ζήτημα του χρέους θα πρέπει να συζητηθεί όπως δεσμευτήκαμε στην αρχή του μνημονίου. Κάποιες φορές ε, παρατηρούμε να οργανώνεται μια, ένας εκβιασμός ε, μεταξύ ενός ή άλλου θεσμού ε, και του τρόπου διεξάγεται η διαπραγμάτευση του χρέους. Και επειδή ουσιαστικά η Ευρώπη ηγείται τις υποθέσεις αυτές, δεν θα έπρεπε η ίδια να στέλνει κάποια μηνύματα ότι έχει φτάσει η στιγμή να ασχοληθούμε ήρεμα με αυτό το ζήτημα και να πει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να κάνει πως δεν ακούει ε, τη θέση αυτής της αντιπροσωπείας που μετέβει εκεί ε, όπως αναφέρετε και εσείς κύριε Αντιπρόεδρε ε, υπό τη δική σας αρχή αλλά και όσον αφορά τη θέση της Κομισιόν. Κοιτάξτε για το χρέος, ας το πούμε. Νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες είναι αντίστροφες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, έχει την αιχμή του δόρατος για το θέμα αυτό. Και άλλωστε αποτελεί και μέρος της συζήτησης. Όσο μεγαλύτερη συνοχή έχουν μεταρρυθμίσεις και όσο ε, πιο ισχυρό το προϊόν των μεταρρυθμίσεων, ε, τόσο λιγότερο φιλόδοξο ε, είναι η παρέμβαση για το χρέος και αντίστροφα. Και γι' αυτό θέλουμε να προσαρμόσουμε τις διάφορες παραμέτρους. Τα δύο θέματα αυτά δεν είναι διαχωριστέα, είναι άρρηκτα δεμένα και πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας στη Ουάσιγκτον θα ξεκινήσουμε να μιλούμε και για τα δύο ε, θέματα μαζί. Όλοι οι δρόντες, οι παράγοντες θα είναι εκεί και θα έχουμε όλες τις παραμέτρους. Θα έχουν ολοκληρώσει τη δουλειά επιτόπου οι επικεφαλής των αποστολών. Θα έχουμε τα δεδομένα, δεν ξέρω να σας πω πόσο θα προχωρήσουμε, αλλά έχει έρθει η στιγμή βεβαίως να συζητήσουμε για το σύνολο. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πίστευω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το μέρος της συνεδρίασης ε, το νόμαδα εργασίας χρηματοδοτικής βοήθειας. Να ευχαριστώ, το, να ευχαριστώ τον Αντίπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τον ε, κύριο Μοσκοβησή. Θα παραμένουμε τώρα για την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Δεν χρειάζομαστε πιστεύω συμπεράσματα. Τα πράγματα είναι σαφή. Υπάρχει μια θετική αξιολόγηση, αναμένουμε θετικό αποτέλεσμα και όλοι ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η έκφραση μέσα στις επόμενες ώρες ή ε, ημέρες. Ας περάσουμε τώρα στον οικονομικό μας διάλογο. όπου θα εστιαστούμε στην διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και την ε, αναθεώρηση που είναι σημαντική ε, γιατί περιλαμβάνει θέματα καινοτομία, ε, αποτελεί καινοτομία και αποτελεί και αξιολόγηση των μακροοικονομικών ισορροπιών ή ανισορροπιών της Ευρωζώνης. Να ζητήσω λοιπόν από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντομπρόφσκης, να παρουσιάσει τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις για το θέμα αυτό και μετά ο Πιέρ ε, συνολικά 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας αυτή στον οικονομικό διάλογο, ο οποίος είναι ουσιώδους σημασίας ε, στη συζήτησή μας για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών συμπεριλαμβανομένων των κοινοτομιών που εισήχθησαν το τελευταίο έτος. Ο Πιέρ στη συνέχεια θα μιλήσει για τις ε, επιμέρους χώρες και περιοχές όπου εντοπίστηκαν ανισορροπίες. Το Φεβρουάριο λοιπόν δημοσιεύσαμε την, ε, σε βάθος ανάλυση για τα 18 κράτη-μέλη που είχαν ε, προσδιοριστεί για περαιτέρω εξέταση στον ε, έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνηση. Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε την αξιολόγησή μα για την Κύπρο, η οποία βγήκε από το τριετέ πρόγραμμα ε, χρηματοδοτική βοήθειας τέλη Μαρτίου και ε, ξαναμπήκε στο τυπικό πλαίσιο συντονισμού οικονομική πολιτική, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Βάσει των αναλύσεών μα, τα κρατημέλη συνεχίζουν να σημαίνουν πρόοδο διορθώνουν τις ανισορροπίες τους, πραγματοποιούνται ε, μεταρρυθμίσεις ε, σε πολλούς τομείς πολιτικής, αλλά η προσπάθεια παραμένει ανομοιόμορφη. Το ίδιο και τα αποτελέσματα. Η προσαρμογή των ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών έχει προχωρήσει, αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί. Ε, υπάρχουν υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημοσίου δανείου, ε, χρέους, συγγνώμη, ή αυξάνονται δυστυχώς σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η ανεργία συνολικά μειώνεται, αλλά παραμένει αρκετά υψηλή σε ορισμένες χώρες, ειδικότερα μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Η ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά το εξωτερικό περιβάλλον ε, ε, έχει, έχει γίνει πιο δυσχερές. Το ίδιο και το πολιτικό πλαίσιο. Ε, τα θέματα ασφαλείας και οι γεωπολιτικές εντάσεις ε, ε, απασχολούν όλους. Η προσφυγική κρίση αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση για όλους τους υπευθύνου χαρακτής πολιτικής στην Ευρώπη και τους υπευθύνου λήψη αποφάσεων. Και είναι σημαντικό να μην υποκύψουμε στην απειλή του λαϊκισμού. Τώρα λοιπόν περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, να απαγιώσει την εμπιστοσύνη και να επιτρέψει οι μεταρρυθμίσει να μετατραπούν σε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία το συντομότερο δυνατόν και στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδο με τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Κοινωνικών Εταίρων και λοιπόν ενδιαφερομένων όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Αυτό απαιτεί ε, ε, δέσμευση και σε βάθος διάλογο. Για να τονώσει αυτή τη διαδικασία η Κομισιόν δημοσίευσε τις εκθέσεις κατά χώρα όπως και το 2015 στις αρχές του έτους. Όπως υποσχεθήκαμε στην ανακοίνωσή μας βήματα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του περσινού Οκτωβρίου, έχουμε επίσης πραγματοποιήσει μια σειρά βημάτων για την ενίσχυση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών και να ενισχύσουμε τη διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή της. Πρώτον, ε, ε, προσδιορίσαμε και απλοποίησαμε τις κατηγορίες ε, του MIP, τις διαδικασίες μακροοικονομικής μακροοικονομικών ισορροπιών, ώστε να υπάρχει ένα πιο απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο και πιο διαφάνες. Οι έξι κατηγορίες λοιπόν των περασμένων ετών μειώθηκαν στις τέσσερις. καμία ανισορροπία, ανισορροπίες, υπερβολικές ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπίες με διορθωτική δράση, δηλαδή με την ε, ε, έναρξη, την ενεργοποίηση της διαδικασίας ε, υπερβολικών ανισορροπιών. Όσον αφορά τώρα τα ευρήματά μας, έξι χώρες διαπιστώθηκε ότι υποφέρουν από υπερβολικές ανισορροπίες. Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Χροατία, Ιταλία και Πορτογαλία και επτά παρουσιάζουν ανισορροπίες. Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία. Ταυτόχρονα τέσσερα κράτη-μέλη που αξιολογήθηκαν βρέθηκαν χωρίς ανισορροπίες Βέλγιο, Ουγγαρία, Ρουμανία και το Νόμονο Βασίλειο και εξήλθαν τις διαδικασίες. Επίσης δεν βρέθηκε καμία ανισορροπία για τις δύο χώρες ε, που υπέστησαν σε βαθμό αναλύση για πρώτη φορά, Αυστρία και Εστονία. Η μείωση του αριθμού των κατηγοριών ε, συνοδεύεται από ισχυρότερη παρακολούθηση Συγκεκριμένη παρακολούθηση στο εξή θα εφαρμόζεται σε όλε τι χώρε ε, στι οποίε έχουν προσδιοριστεί ανισορροπίε. Φυσικά θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα των ανισορροπιών που υφίστανται οι χώρε. Δεύτερον, παρουσιάσαμε τα ευρήματα κάθε ε, σε βαθμό αξιολόγηση με τη βοήθεια ενό πίνακα αξιολόγηση ε, MIP διασφαλίζοντα την σαφή και διαφανή τη παρουσίαση. Τέλος, ε, σύντομα θα δημοσιεύσουμε ένα εγχειρίδιο του MIP που θα παρουσιάζει τη νομική βάση του MIP, θα διευκρινίσει τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τις αναλύσεις της Κομισιόν και θα, ε, θα παρουσιάζει ένα απολογισμό της υλοποίηση ε, στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας. Όλα αυτά τα βήματα βοηθούν να βελτιωθεί η διαφάνεια και η σαφήνεια στον τρόπο υλοποίηση του MIP και θα το ενισχύσει ως εργαλείο επιτήρησης και συντονισμού πολιτικής. Ο Πιέρ τώρα θα σας παρουσιάσει τις συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις ε, για συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Παλτής, λέει ο κ. Μοσκοβισή. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για εντατικοποίηση διαχείριση εξωτερικών κινδύνων, χρειάζεται ε, νέα εξισορρόπηση των οικονομιών ε, και στην Ευρωζώνη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έλεγα με δύο λόγια για την έκθεση του 2016. Πιο ε, λεπτομερώς θα ήθελα να σας πω ότι 16 χώρες ήταν ήδη σε επιτήρηση για τα μακροοικονομικά θέματα. Δεν θα υπενθυμίσω τον κατάλογο. Έγινε εις βάθος ανάλυση για την Αυστρία και την Εστονία για πρώτη φορά ε, ε, μετά την ε, έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπης του Νοεμβρίου 2015. Επίσης έγινε ένας απολογισμός για την Κύπρο. 19 χώρες έχουμε στη διαδικασία τελικά. Τονίζω τα οριζόντια θέματα που προκύπτουν από αυτή τη δέσμη απολογισμών και εκθέσεων. Καταρχήν, συνεχίζουν οι οικονομικές προκλήσεις ε, σε πολλές περιπτώσεις τα ελλείμματα μετατράπησαν σε πλεονάσματα και θα πρέπει να συνεχίσουν ορισμένες χώρες αυτή την κατάσταση ε, πλεονασμάτων. Η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή έχει ένα από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα του κόσμου. Υπάρχουν βεβαίως Κάποιε διαφοροποίησει οι οποίε βρίσκονται να εξελίξει. Ε, υψηλό επίπεδο χρέου είναι άλλο ένα οριζόντιο ζήτημα που παραμένει ανησυχητικό. Είναι ιστορικά υψηλά τα επίπεδα χρέου σε πολλέ χώρες και σε πολλούς τομεί της οικονομία ε, των νοικοκυριών ε, μεταξύ άλλων. Παραμένουν δυσκολίες λοιπόν προς επίλυση. Περνώ τώρα ε, στις ε, εμπεριστατωμένες εκθέσεις. Έξι χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, ε, Πορτογαλία και Κύπρος έχουν μακροοικονομικές, εξαιρετικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Κύπρος πρώτη φορά μπαίνει στη διαδικασία αυτή μετά την πρόσφατη εξοδότηση από το πρόγραμμα βοήθειας και θα ξαναμπεί άμεσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Για τις άλλες πέντε χώρες θα έλεγα ότι ε, κρατάμε την ε, ίδια κατηγοριοποίηση η διαδικασία διόρθωσης παραμένει μία από τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις και η Επιτροπή θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Επτά χώρες έχουν κατάσταση ανισορροπίας. Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Φινλανδία, Σλοβενία και Σουηδία. Αυτό είχε επισημανθεί και πέρυσι για τις χώρες αυτές, αλλά έχει μειωθεί ο ρυθμός των κατηγοριών, όπως είπαμε πριν, για να μπορέσει η διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική. Τέλος, για έξι χώρες φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανισορροπία. Βέλγιο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και δύο χώρες για τις οποίες έγινε για πρώτη φορά εμπεριστατωμένη έκθεση Αυστρία και Σλοβενία. Τώρα για τα επόμενα βήματα θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή ε, θα συνεχίσει να εξετάζει τα προγράμματα σταθερότητας που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη και τα προγράμματα σύγκλησης και σταθερότητας που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη και θα εκδοθούν στις αρχές Μαΐου. Το Μάιο επίσης η Επιτροπή θα συντάξει τις ειδικέ ε, συστάσεις αναχώρα και ορισμένε από τις συστάσεις αυτές ε, θα αποσκοπούν στη διόρθωση των ανισορροπιών που εντοπίστηκαν κατά τις εμπεριστατωμένες εκθέσεις. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Παύλο Ζάλμπερ είναι πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης και Επίτροπε Μοσκοβισή, σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας ε, δώσατε σήμερα. Θα μιλήσω για τη χώρα μου, την Ισπανία, η οποία δεν ε, πέτυχε το στόχο του ελλείμματος και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο λόγω του ότι οι αυτόνομες κοινότητες, οι ισπανικές περιφέρειες δεν τήρησαν τους στόχους τους επιμέρους του ελλείμματος. Και ε, είμαστε δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και έχουν ανακοινωθεί μέτρα για καλύτερο έλεγχο των δημοσίων δαπανών στις περιφέρειες στις περιφέρειες, στις αυτόνομες κοινότητες. Και ο σχετικός νόμος έχει εφαρμοστεί με αρκετά και πολλά σκληρά μέτρα. Είχαμε έλλειμμα 9% και καταφέραμε να το μειώσουμε ε, στο μισό Έχουμε λοιπόν διανύσει μεγάλη απόσταση. Θα ήθελα να κάνω ανάλυση της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Δύο είναι οι πιθανότητες. Ένας μεγάλος κυβερνητικός συνασπισμός ή μια κυβέρνηση στην οποία να συμμετάσχουν τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν θα σας ζητήσω να μας πείτε ποιο προτιμάτε βεβαίως από τα δύο, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να αξιολογήσετε ορισμένες προτάσεις που συζητούνται, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια να εξαιρεθούν, να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες ή να αναδιαρθρωθεί το δημόσιο χρέος. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικών δυσκολιών είναι συμβατές αυτές οι δυσκολίες με τέτοιου είδους πολιτικές που θα επιφέρουν αύξηση δημοσίων δαπανών και θεωρείται ότι είναι συμβατό να ε, μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης εάν τελικά η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, ε, αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες και ε, κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Απάντηση. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Ακούγοντάς σας όμως χαμογελώ κάπως, διότι ε, ε, σκεφτόμαι το παρελθόν. Όταν παρουσίασα μία άποψη ε, που ε, έπρεπε από το 4,7 στο έλλειμμα να πάμε στο 4,2 ε, στο έλλειμμα στην Ισπανία η υποδοχή του που μου επιφύλαξε ο Ισπανικός τύπος ήταν αρκετά οδυνηρή Τώρα Θέλω να πω με αυτά ε, και ε, ότι πράγματι μπορούν να γίνουν προσπάθειες και η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντείνει ε, προς αυτή την κατεύθυνση εξού και άλλωστε το έλλειμμά σας τώρα είναι στο γύρω στο 5%. Μπορώ να απαντήσω εμέσως στο ερώτημά σας. Όποια και αν είναι η κυβέρνηση και επαναλαμβάνω όποια και αν είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να επανέλθουμε στο πλαίσιο των απαιτήσεων που είναι κοινέ για όλους στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Τώρα, ε, με, με διάφορες προθεσμίες βεβαίως το, ε, είναι το θέμα στο τραπέζι και ότι ο κύριος Ραχώε είχε ζητήσει προθεσμία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις ευθύνες της και θα αξιολογήσει το κατά πόσο η κάθε χώρα τηρεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Το κάνει αυτό η Επιτροπή και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Θα συνεχίσει να το κάνει. Ο Πρόεδρος. Να προσθέσω δύο λόγια στα λεγόμενα του Πιέχ Πράγματι, το Μάρτιο δημοσιεύτηκαν ξεχωριστές συστάσεις για την Ισπανία οι οποίοι στάθηκαν ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, στον έλεγχο των δαπανών σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό ήταν το βασικό στοιχείο ε, για το, ε, λόγω του οποίου η Ισπανία απόκλινε του δημοσιονομικού τους τη στόχου πέρσι. Και αυτό είναι αυτό ε, για το οποίο συζητούμε με τις ισπανικές αρχές. Πώς θα υπάρξει δημοσιονομική ε, πειθαρχία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Για να ε, έχουμε ε, συνολική ισορροπία δημοσιονομική σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης. Αυτό είναι σαφέστατο. Τώρα, επιπρόσθετα βήματα μπορεί να γίνουν μαζί με την αξιολόγηση που θα έχουμε για τις άλλες χώρες τον Μάιο, έχοντας λάβει τα δεδομένα τα οποία θα έχει επικυρώσει η Eurostat και έχοντας διαβάσει τη δημοσίευση για τις οικονομικές προβλέψεις της ΕΑΡΙΝΕΣ που θα επικαιροποιούν και θα ενημερώνουν τα δεδομένα μας. Το Μάιο λοιπόν θα επανέλθουμε στην εξέταση ανα περίπτωση αναχώρα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Και ε, για ορισμένες χώρες θα εξετάσουμε και την τήρηση του στόχου ε, ε, δηλαδή του Συμφώνου Σταθερότητας. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμπλέκεται στις κομματικές πολιτικές, ε, στο κομματικό και πολιτικό γίγνεσθε μέσα στις χώρες. Αυτό είναι σαφέστατο. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η Ισπανία έχει κάνει πολύ σημαντικές προόδους. Ε, έχει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη με μέσο όρο ανώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ και η ανεργία αυτή τη στιγμή ε, είναι σε καθολική πορεία παρόλο που παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όλα αυτά είναι καλά λοιπόν και το σημαντικό είναι να μην παρεκκλίνει η Ισπανία από την τροχιά για να μην υπονομευθεί η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και ως προς το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι σημαντικό να μην δημιουργείται αβεβαιότητα. Η Ισπανία είναι απολύτως σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε καν να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το momentum την ορμή και να μην απολεστεί η εμπιστοσύνη των αγορών σε σχέση με τη δυνατότητα της Ισπανίας να χρηματοδοτεί και να χρηματοδοτεί το χρέος της με λογικά επιτόπια. Ε, λέει ο κύριος Δομπρόφσκης. Ευχαριστούμε πολύ. Ελίζα Φερέιρα. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να αναφερθώ στην ισπανική περίπτωση, αλλά αφού το ανέφερε ο Παύλο, Φυσικά όλοι μας ε, έχουμε στραφεί με μεγάλη προσοχή προς την Κομισιόν και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα οι προσπάθειες που ζητάτε από τα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί πάντα υπάρχει έτσι, προσπαθεί κανείς να καταλάβει την ορθότητα, την ισορροπία, το πόσο σωστή ε, θα είναι και ισόρροπη η εφαρμογή της νομοθεσίας. Αλλά ίσως να μην είναι το θέμα που πρέπει να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή αυτό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να διασφαλίσει τη συμμορφώση με τους κανόνες ε, έλαβε μια επιστολή από 7 υπουργού οικονομικών ή ε, κομισιών, ε, μέσα τη οποία ζητείται κάποια προσαρμογή λογική, φαίνεται, ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την επιτύχηση τη ισορροπία. Έχετε ασχοληθεί με αυτό, γιατί η διαρθρωτική ισορροπία φαίνεται ότι είναι ένα, κάτι, κάτι σαφές που δεν καταλαβαίνει κανείς, οπότε Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να δούμε πώς μπορούμε να δούμε με τον ίδιο τρόπο αυτές τις τιμές, όλα αυτά τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία. Τώρα το ερώτημά μου αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει. Η Κομισιόν αντιμετωπίζει και σας συγχαίρω τον τρόπο με τον οποίο ε, φέρνουν αποτελέσματα αυτά τα εργαλεία, όλα αυτά τα μέσα, οι μηχανισμοί. Ωστόσο η Κομισιόν συνεχίζει να επαναλαμβάνει την ίδια ανάλυση υπερβολικών ε, ελλημάτων ε, επικεντρωνόμενη στις μακροοικονομικές μεταβλητές κατά τη χρήση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπίων ενώ αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε ε, τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας ε, και ποιες είναι οι συνέπειες. Οπότε η ερώτησή μου είναι, αν δούμε τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα σχετικά εθνικά προγράμματα, σκοπεύετε να βγείτε από αυτό το σκεπτικό της συμμόρφωσης και της μη συμμόρφωσης και να δείξετε ότι είστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι, ότι μπορείτε να καταλάβετε την πραγματική κατάσταση των οικονομιών. Θα τελειώσω ένα λεπτό. Ε, όχι, λέει ο Πρόεδρος. Απλά να πω 20 από τα 28 κράτη-μέλη έχασαν ε, μερίδια αγορά ε, στον τομέα των εξαγωγών τελευταία πενταετία. Ωραία, λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για την επιστολή των Υπουργών Οικονομικών των 8 κρατών μελών η οποία αφορούσε το χρονικό οριζόντα και το κενό των επιδόσεων όσον αφορά τις προβλέψεις της Κομισιόν. Ε, το μελετάμε αυτή τη στιγμή με μεγάλη προσοχή. Ε, εξετάζουμε τις επιπτώσεις και εγώ πρόσφατα μίλησα με τον Υπουργό Οικονομικών της Ιταλίας, τον Πιερ Καλοβαδόν, που προφανώς ηγείται αυτής της άσκησης. Σημειώθηκε όμως ότι αυτή είναι μια κοινά συμφωνηθής μεθοδολογία Δηλαδή έχει συμφωνηθεί και από τα 28 κράτη-μέλη και πρέπει επίσης να συμφωνούνται και οι τροπολογίες, οι τροποποίησεις σε αυτήν από όλα τα κράτη-μέλη και τα 28. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση ε, θα υπάρξει συζήτηση στην ομάδα εργασίας ε, Output Gap, όπως λέγεται, για να βρεθούν ε, οι κατάλληλες ε, λύσεις. Όπως γνωρίζετε αυτά τα κενά αποδόσεων ε, είναι πολύ περίπλοκα. Ε, δεν είναι υπολογισμοί που μπορούν να εξηγηθούν εύκολα. Και στη δική μας προσέγγιση τώρα ε, προσπαθούμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εξετάζουμε το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα του παραγωγικού χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο απλούς δείκτες και αποτελεσματικούς. Αξιολογούμε λοιπόν αυτό το αίτημα ανοιχτό μυαλά, αλλά η Κομισιόν δεν μπορεί να το αλλάξει μονομερός διότι είναι κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί ως μεθοδολογία από κοινού και από τα 28 κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, όπως γνωρίζετε υπάρχει ένας ε, πίνακας βαθμολογίας βάσει δικτών, ε, βάσει το οποίο κάνουμε τις αξιολογήσεις των ε, οικονομιών των κρατών μελών και έτσι προκύπτουν οι συστάσεις κατά χώρα. Να πω ότι Συχνά αυτές οι στάσεις είναι ποιοτική φύσης, ε, όχι πάντα ποσοτικές. Πρόκειται λοιπόν για μια ποιοτική αξιολόγηση της οικονομίας ενός κράτους μέλους, ε, όπου αναφέρονται οι βασικοί τομεί όπου απαιτούνται βασικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθούν οι οικονομικές επιδόσεις σε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο. Τώρα δεν ξέρω, ο Πιέρ θα θέλει να απαντήσει. Δύο λόγια. Οι χώρε αυτές σαφώ ε, και θα είναι στο επίκεντρο τη προσοχής μας και με μεγάλη προσοχή θα εξετάσουμε αυτά τα στοιχεία. Θα περάσει και από το Eurogroup. Και όσον αφορά την τρέχουσα διαδικασία θα γίνει με τους υφιστάμενους κανόνες. δεύτερη παρατήρηση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η εμπεριστατωμένη ανάλυση μας αφορούσε όλους τους παράγοντες. Και μαζί με τον Βάλτης Ντομπρόφσκης προσπαθούμε να βελτιώσουμε ποιοτικά αναχώρα ε, της αναλύσης Thank Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι εγώ θυμάμαι διαφορετικά τα θέματα της, των προοπτικών και του παραγωγικού χάσματος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε ε, αυτά που μας φανεί η Επίτροπη. Ο Μπέρντ Λούκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη. Διάβασα την έκθεση για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και κάτι το οποίο δεν βρίσκω είναι μια βασική ανισορροπία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ανισορροπία στην αγορά κεφαλαίων δηλαδή. Είναι η τόκη γύρω στο μηδέν και αρνητική θα έλεγα. Πολύ μικρή ζήτηση πιστώσεων και οι αποφάσεις ε, των πολιτών για αποταμίευση είναι πάρα πολύ ε, χαμηλές ε, και γίνεται και πιο δύσκολη η διαδικασία ανάληψης των δαπανών για τον γυράσκοντα πληθυσμό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη μακροοικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ένα τόσο βασικό παράγοντα όπως είναι τα επιτόκια. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρετε αυτά τα πολύ χαμηλά έως και αρνητικά επιτόκια όταν μιλάτε για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν θέλετε να εκφέρετε καμία κριτική για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρείτε ότι είναι υπεύθυνη η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα. Διαφωνείτε με ε, τις γερμανικές απόψεις που έχουν ακουστεί από τον ε, Υπουργό σχετικά με αυτό το θέμα. Πρόεδρος, νομίζω ότι ήταν ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Ντομπρόφσκης. Όντως, όσον αφορά την ε, νομισματική πολιτική, νομισματική πολιτική είναι κάτι ε, το οποίο καθορίζει με ανεξάρτητο τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμβουλεύει. την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε δίνει σχετικές εντολές. Γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει χαμηλός και μερικές φορές είναι και αρνητικός και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο χαμηλά από τον στόχο πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας που είναι κάτω από το 2%. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ποσοτική ελάφρυνση, για την ποιοτική ε, ελάφρυνση κλπ. λαμβάνονται με στόχο να επιτευχθούν ή ο στόχος πληθωρισμού που έχει θέσει η ο στόχος πληθωρισμού που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τα χαμηλά επιτόκια, ή τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την κλασική νομισματική πολιτική, βαίνουν αντίθετα, δηλαδή ακριβώς αυτό κάνει και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βρισκόμαστε στα όρια βέβαια αυτής της πολιτικής και οι παρενέργειες της πολιτικής αυτής εμφανίζονται στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Όντως ισχύει αυτό και είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε. Όσον αφορά ε, την προσφορά και ζήτηση στον πιστωτικό τομέα, εδώ υπάρχουν πολλές ε, δίσταμες απόψεις. Οι τράπεζες λένε ότι δεν υπάρχει ζήτηση, οι επιχειρήσεις, ιδίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λένε ότι δεν υπάρχει προσφορά. Ίσως κάπου στη μέση λοιπόν να βρίσκεται η αλήθεια. Όμως, ε, όντως, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να καταλήγει σε περισσότερες πιστώσεις για την πραγματική οικονομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους για να το επιτύχει αυτό, όχι μόνο μέσω των τραπεζών αλλά και μέσω των κεφαλαίων και γι' αυτό υπάρχει και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση κεφαλή αγορών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζουμε πάντοτε και εμείς και ο κύριος Δράγκη. Μόνο με την νομισματική πολιτική δεν μπορούν να επιληθούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν επικοδομητικά το χρόνο τους ε, για να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να βοηθήσουν την οικονομία τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να τους αφήσει κάποιο χρονικό διάστημα για να το επιτύχουν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει εν σοφία να χρησιμοποιήσουν αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Ενρίκε Καλβέ ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κύριε Επίτροπε. Με λακωνικό τρόπο θα προσπαθήσω να απευθύνω όλες μου τις ερωτήσεις σε εσάς. Πρώτον, είναι κάπως ε, ιδιωτεύον με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου να προσπαθεί κανείς να βελτιώνει τα MIP. Ε, στερούνται ευρωπαϊκού οράματος, να δούμε το σύνολο και όχι διαφοροποιημένα τι γίνεται σε κάθε χώρα, γιατί έτσι γίνονται τα μέτρα εξαιρετικά εθνικιστικά. Πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκή ισορροπία σε μια ύπρο που θα πρέπει να προχωρά προς περισσότερη ισότητα. Δεύτερον, η αντιμετώπιση κάθε έθνους πρέπει να είναι ίδια για όλους και ε, τα, οι ανισορροπίες οι πλεονασματικές δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις ελληματικές ανισορροπίες και άλλοι είναι η μεταχείριση της Γερμανία και άλλοι της Πορτογαλίας και αυτό είναι με πάσα ειλικρινία πολύ κακό εάν ε, ε, θέλουμε να διατηρήσουμε τα πλεονάσματα, αυτό είναι πολύ καλό. Και αν θέλουμε να δείξουμε παραδείγματα μικρών χωρών που δεν ενοχλούν, όλα αυτά είναι πολύ ε, ε, κακά. Υπάρχει αίσθηση αδικίας και άνησης ε, μεταχείρισης και διαφορετικής μεταχείρισης και γι' αυτό τελικά δεν υιοθετούνται από τα κράτη τα σωστά μέτρα. Η Πορτογαλία έκανε όλα τα μαθήματα άριστα και αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση ε, εκ του επιτήρησης. Δεν θα δουλέψει. Ό,τι και να ζητάτε δεν θα δουλέψει αν δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική επιθετική ε, στο φορολογικό επίπεδο για να, στο δημοσιονομικό επίπεδο μάλλον, για να αντισταθμίσουμε αυτό που γίνεται ε, στο νομισματικό επίπεδο. Πού έχει πάει αυτή η ιδέα για ένα fiscal board για όλη την Ευρώπη. Και θα ήθελα να μιλήσω τώρα στα Ισπανικά, γιατί θα μιλήσω για τη χώρα στην οποία εκλέγομαι, την Ισπανία. Ε, πολύ σύντομα ε, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό ε, θα μπούμε ως Ισπανία σε χώρα στενής παρακολούθησης, σε κατάσταση στενής παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό το 25% θα υπάρξουν πρόστιμα ε, εν πάση περιπτώσει παρατείνεται ε, ε, κατά ένα χρόνο γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε τόσα λεφτά από το μανίκι μας. Σε κάθε περίπτωση στην Ισπανία δεν μπορούμε να πληρώνουμε αυτό το σύστημα το οποίο δεν μπορεί να το κυβερνήσει κανείς της επιβολικής περιφερειοποίησης και ύπαρξης αυτόνομων κοινοτήτων και τόσο μεγάλης αυτονομίας γενικότερα. Ευχαριστώ. Απάντηση του κυρίου Μοσκοβισή. Ως προς τη διαδικασία MIP γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αναγκαιότητά της, να γίνει πιο ευανάγνωστη αν θέλετε από το κοινό, από την κοινή γνώμη. Και γι' αυτό έχουμε ενισχύσει την επιτήρηση και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε μια προσέγγιση πιο συνολική του συνόλου των προβλημάτων. Τώρα, ως προς τις εκτιμήσεις σας, για το πώς λαμβάνονται υπόψη τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα, συμφωνώ μαζί σας. Δεν πρέπει να υπάρχει ανισότητα στην εκτίμηση μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το στάδιο έχουμε ταξινομήσεις και κατατάξεις οι οποίες είναι έγκυρες. Λίγες είναι οι αλλαγές από τη μία χρονιά στην άλλη. Ε, θεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρέπει να προχωρήσει παραπάνω αυτή η διαδικασία στις περιπτώσεις που το θεώρησε. Ωστόσο, οι χώρες με μεγάλα πλεονεάσματα πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουν τα υπερβολικά πλεονάσματα. Βέβαια αναφέρομαι σε όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ε, προσφυγική κρίση που θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο και θα πρέπει και αυτός να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου. Τώρα, ε, για το Fiscal Board, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχουν υπάρξει συνεδριάσεις, υπήρξε απόφαση τον Οκτώβριο. Είναι ένας παράγοντας περισσότερης Ευρώπης, αυτό ε, είναι σίγουρο. Τώρα για την Ισπανία να ξαναπώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε χρήσιμο χρόνο, σε έφθετο χρόνο, τον Μάιο, θα υιοθετήσει ε, τις απαραίτητες διατάξεις. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Μιγγέλ Πιέγας. Ε, particular a ε, parte sobre ε, Portugal. Διάβασα την έκθεση και ειδικότερα το κομμάτι για την Πορτογαλία και αυτό που διαφαίνεται αντικειμενικά είναι η αποτυχία ολόκληρης της στρατηγικής στην οποία βασίστηκε η παρέμβαση της Τρόικα η χώρα δεν γνώρισε ανάπτυξη, λέγεται και στην έκθεση. Οι δυνατότητε ανάπτυξη είναι χαμηλέ, μειώθηκαν οι επενδύσει, αυξήθηκε η ενεργεία. Χάσαμε δεκάδες χιλιάδες ε, νέους εξειδικευμένους που έφυγαν από την Πορτογαλία, ερευνητέ, για παράδειγμα, γεγονός ε, που δυσχεραίνει το μέλλον και την οικονομική ανάπτυξη της Πορτογαλίας. Αλλά υπάρχει και κάτι καινούριο. Τώρα είχαμε εκλογέ στην Πορτογαλία και ο Πορτογαλικό λαός απέρριψε τις πολιτικές αυτέ. Απέρριψε αυτή την δημοσιονομική μεταρρύθμιση που οδήγησε σε αύξηση των φόρων για τους εργαζομένους και σε μείωση των φόρων για τις επιχειρήσεις. Ο κόσμος, ο λαός απέρριψε όλες αυτές τις δυνατότητες ε, όλες αυτά τα μέτρα για την αγορά εργασία, διότι δεν, υπήρξε, δεν έφεραν αποτέλεσμα, αύξησαν τη φτώχεια, δεν επέλυσαν τα προβλήματα των δημοσίων οικονομικών όπω αναγνωρίζεται και στην έκθεση την ίδια. Το πρόβλημα τώρα λοιπόν έχει ως εξή. Τι μπορεί να κάνει κανεί υπό αυτέ τι περιστάσει. Πώ μπορείτε να επιμένετε στι ίδιε πολιτικέ οι οποίε έχουν αποτύχει και επιπλέον απορρίφθηκαν από του ψηφοφόρου, από ε, τη λαϊκή φωνή. Εάν στην παρούσα φάση δεν καταφέρουμε να βρούμε εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αντιστρέψουν, να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο ύφεση και εξάρτησης, εάν δεν βρούμε μέτρα αύξησης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την υποστήριξη της κατανάλωσης, εάν δεν να, το δημόσιο χρέος, ε, πρόβλημα παγκόσμιο, όχι μόνο της Πορτογαλίας, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα και να το επιλύσουμε. Δύο λεπτά ακριβώ, λέει ο πρόεδρο. Ε, ε, περισσότερη πειθαρχία δείξατε από άλλου. Ε, θα είμαι και εγώ το ίδιο σύντομο. Να πω απλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και στην περίπτωση της ε, Ισπανίας, δεν πρόκειται να αναμειχθεί στην στον πολιτικό βίο της Πορτογαλίας. Δείχνουμε κάποιο σεβασμό. Είχαμε κάποια ανταλλαγή με την Πορτογαλική κυβέρνηση βάσει τις οποίες αποφύγαμε, το οποίο αποτελούσε κοινό στόχο, την απορρίψη του προσχεδίου του προπολογισμού και λήφθησαν μέτρα τα οποία επέτρεψαν να παραμείνουμε εντό των αποδεκτών περιθωριών μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματο. Και όλα αυτά έγιναν σε πολύ καλή συνεννόηση με την Πορτογαλική κυβέρνηση εξαιρετικά εύκολα. Ήταν πολύ γρήγορε και εύκολε συζητήσει ε, και από τι δύο πλευρέ. Εγώ ίδιο ε, στη συνέχεια μετέμεινε στη Λισαβόνα ε, πιστεύω ότι τα μηνύματα που ανταλλάξαμε ήταν θετικά. Ο Πρωθυπουργό Αντώνιο Κώστα μόλι εχθέ ε, ε, διευκρίνησε τι θα κάνουμε, πώ θα αντιμετωπίσουμε πάντω είδου ενδεχόμενα και σενάρια. Και έτσι υπάρχει μια συνεννόηση με την Πορτογαλική κυβέρνηση για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση εντό του χρονοδιαγράμματο που έχει προβλεφθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να παρουσιάζουμε τα πράγματα με δραματικό τρόπο, ούτε να συμπεριφερόμαστε ανταγωνιστικά. Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Πορτογαλίας ε, είναι πολύ υψηλή ποιότητα και πιστεύω ότι αυτό έχει αναγνωριστεί από άπαντε. Ευχαριστώ. Ernest Τρεις σύντομες ερωτήσεις. Στην έκθεση μιλάτε για την βιωσιμότητα των δημοσίων λογαριασμών και τη δυνατότητα ανάκαμψης και ανάκτησης των οικονομικών δεδομένων. Στην Ισπανία έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης ε, μεγαλύτερος από το μέσο όρο, αλλά οφείλεται σε πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Μήπως ε, δουλεύετε με εξαιρετικά μειωμένους ε, πολλαπλασιαστές, υπάρχει συμπέρασμα γι' αυτό. Και το λέω αυτό δεδομένου ότι δεν μας προσέχουν οι σε αυτή τη στιγμή και άρα μήπως έχουμε περισσότερο χρόνο για να φύγουμε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και δεν μας δίδεται. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ο συνάδελφος από το ΕΛΚΕ μιλάει για τις ευθύνες των αυτόνομων κοινοτήτων, οι οποίες όμως διαχειρίζονται μόνο το 1 τρίτο των ε, ελλημάτων και τελικά ευθύνονται μόνο για το 1 έκτο του ελλείμματος που επιτρέπεται. Είναι δύο βασικοί κίνδυνοι να μην τηρηθεί το όριο του ελλείμματος σε σχέση με ε, τα έσοδα τις, τα ασφαλιστικά αλλά και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα κάνετε ανεξάρτητες μελέτες για να βρείτε πού ακριβώς είναι το πρόβλημα ή θα λέτε όπως το Λαϊκό Κόμμα ότι την ευθύνη την έχουν οι φορείς της κυβέρνησης που ε, βρίσκονται στις αυτόνομες κοινότητες μόνο θα ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις για την προσαρμογή του ελλείμματος με την προσωρινή κυβέρνηση ή θα περιμένετε ε, να προκύψει δημοκρατικός νομοποιημένη εκλεγμένη νέα κυβέρνηση για να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ο κ. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ισπανία, όπως ε, ήδη είπαμε, είναι περίπλοκη η κατάσταση. Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βλέπουμε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για την οικονομική ανάπτυξη είναι πάνω από το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης φαίνεται τα τελευταία χρόνια βελτίωση Επομένως, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι παράγουν αποτελέσματα. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, έχουμε προκαταρκτικά δεδομένα που μας έχουν δώσει οι Ισπανικές αρχές που δείχνουν ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα ήταν αυτό που αφορούσε τις περιφέρειες. Θα αναλύσουμε τα στοιχεία αφού τα επαληθεύσει η Eurostat και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Και μετά την επαλήθευση της Eurostat αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιήσουμε για τη λήψη αποφάσεων. Όπως ε, είπαμε και πάλι όμως, Το θέμα του ελέγχου των ελλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στις συστάσεις τις οποίες ε, στείλαμε προς την Ισπανία. Για την ερώτησή σας αν θα διαπραγματευτούμε με την τωρινή κυβέρνηση, αν θα περιμένουμε την ε, νέα κυβέρνηση, έχουμε ξαναπεί ότι η διαδικασία εκλογών δεν ε, θα έπρεπε να εμποδίζει μια χώρα από το να ακολουθεί τους δημοσιονομικούς και μαρκοοικονομικούς κανόνες. Αναμένουμε λοιπόν από την Ισπανία ε, να ακολουθήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεών της όπως και οποιαδήποτε άλλη χώρα και συζητάμε και με την ε, τρέχουσα κυβέρνηση που ασκεί τα καθήκοντα αυτή τη στιγμή περιμένοντας τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Μπερνά Μονό. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η διαδικασία εμπεριστατωμένων εκθέσεων ανακράτως μέλος θεωρώ ότι είναι αναποτελεσματική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ακατανόητη αυτή η διαδικασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι εντελώς αναποτελεσματική. Η η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το ίμιση των εκθέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Είναι εσφαλμένοι οι στόχοι της Επιτροπής. Αντί να ασχολείται με τη διαχείριση σε κάθε κρατός μέλος, θα πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή τις πραγματικές μακροοικονομικές ανισορροπίες και το γερμανικό ισοζύγιο πληρωμών. Με το εννέο νόμισμα με τις ε, ανταλλαγές μεταξύ κρατών, ε, ασχολήθηκε με τις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αλλά ε, θα πρέπει να μην αγνοείτε τις χώρες οι οποίες κατατρώγονται από τα μεγάλα πλεονάσματα ορισμένων χωρών και ένα το παράδειγμα είναι η μεγάλη λιτότητα στην Ελλάδα. Ακόμη και η Αμερικανική κυβέρνηση στο G20 ζητά να μειωθεί το γερμανικό πλεόνασμα. Το πραγματικό θέμα για να ξαναρχίσει η παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας ε, είναι να ρυθμιστεί το πρόβλημα αυτό των πλεονασμάτων της Γερμανίας. Αλλά ο Γερμανός Υπουργός αγνοεί αυτές τις παρενέσεις και συνεχίζει η Γερμανία να εξάγει ύφεση σε όλες τις χώρες μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δράματα. Εναλλακτική λύση θα ήταν να δρούμε σε μια κοινή νομισματική ζώνη όπου τα κράτη μειώνουν τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα έπρεπε η Επιτροπή αναχώρα να εξετάσει το επίπεδο επαγρύπνησης για να μπορεί να διορθώνει αναχώρα τις ανισορροπίες. Ευχαριστώ. Ο κ. Μοσκοβηθή. Ε, δεν ε, θέλω να ε, κρίνω ρητορικά τα ερωτήματά σας. Θα πρέπει να παραβλέψω αυτά που είπατε για την αναποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ασχοληθώ ε, πιο σοβαρά με την ερώτησή σας και όχι μόνο με τα ρητορικά τεχνάσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως φροντίζει για τη λειτουργία της Ευρωζώνης, κάτι το οποίο ε, προτιμούν οι Ευρωπαίοι, ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει σε όσους διαφωνούν με αυτή τη θέση θέλουμε να έχουμε μια έξυπνη ανάγνωση του Συμφώνου Σταθερότητας προσπαθώντας να έχουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις επιτρέπουν να βελτιώσουμε την συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και προσπαθούμε και να επιλύσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Σε αυτό το θέμα ίσως δεν κατάλαβα επαρκώς το ερώτημά σας, γιατί νομίζω ότι ακριβώς αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Αν υπάρχουν πολλές κατηγορίες, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ανταποκριθούμε στις διάφορες ανισορροπίες. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις συστάσεις μας και γι' αυτό και προσπαθούμε συνεχώς να τις βελτιώνουμε και προσπαθούμε να είναι περισσότερο σφαιρικές, περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα και προσπαθούμε να έχουμε συνεχώς διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κύριε Μονό, προσπαθείτε Ματέως να αποδείξετε το ίδιο πράγμα πάντοτε. Το ευρώ είναι κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι καλό που θέλετε μια σφαιρική και παγκόσμια προσέγγιση από τη μια πλευρά, γιατί καταλήφθηκε το επιχείρημά σας αφετέρου. Ο κύριος Μονό. Μπορώ να δευτερολογήσω κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε το χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος, ο Βαντεν Κεντελάρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά. Όλο επαναρχόμαστε στο ίδιο σημείο φοβάμαι. Είναι σαν να χτυπάτε με ένα σφυρί το ίδιο καρφί, αλλά το καρφί να μην καρφώνεται, αλλά να το χρειαζόμαστε για να στηρίξει όλο τον οίκο μας μόνο 4% όλων των συστάσεων έχουν υλοποιηθεί και έξι χώρες ε, αναφέρθηκαν αλλά η Κομισιόν ε, δεν θέλει να διορθώσει το MIP τώρα και το Συμβούλιο και άλλοι έχουν πει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το MIP σωστά Γιατί λοιπόν η Κομισιόν δεν έχει ακόμα αποφασίσει να ξεκινήσει διαδικασίες μακροοικονομικών ανισορροπιών. Είναι επειδή δεν είναι δυνατόν. Και αν δεν είναι δυνατές χρειάζεται κάποια ενίσχυση διαδικασία, χρειάζεται κάποια μεταρρύθμιση, ε, κάποιες νέες ε, αλλαγμένες συμφωνίες που πρέπει να συνάψουμε με τα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για την υλοποίηση των συστάσεων ε, αναχώρα, να ζητήσω συγγνώμη, μιλήσατε πολύ γρήγορα, οπότε δεν ξέρω αν πρόλαβε ο Δερμηνέας ε, να το αποτυπώσει ακριβώ. Στην αγγλική μετάφραση άκουσα 4% ε, υλοποίηση των συστάσεων. Να αμφισβητήσω λίγο αυτά τα νούμερα. Ακόμα μελετάμε τα φετινά νούμερα, αλλά τα περσινά νούμερα έδειξαν ότι αν μετρήσουμε τις συστάσεις που πλήρως υλοποιήθηκαν, τότε αυτές αντιστοιχούν στο 10% περίπου. Αν λάβουμε επιπλέον υπόψη τα διάφορα, την υλοποίηση, τη μερική υλοποίηση σε διάφορα στάδια, οδηγούμαστε σε ένα 40%. Φυσικά το 40% σε θέματα υλοποίηση δεν είναι κάτι που μα κάνει περήφανου. Συνεπώ απαιτούνται και περαιτέρω προσπάθειε για να βελτιωθεί η υλοποίηση. Και πιστεύω ότι ο πρωταρχικό στόχο θα είναι να ενισχύσουμε την αίσθηση οικειοποίηση ιδιοκτησία των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμένου συμπεριλαμβανομένου του να κάνουμε την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θέμα συζήτηση στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν πέρσι αλλάξαμε το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δημοσιεύονται οι εκθέσεις αναχώρα νωρίτερα, ακριβώς ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και εντός των κρατών μελών, δηλαδή όχι μόνο με τις κυβερνήσεις, αλλά και με τα κοινοβούλια, του κοινωνικού εταίρους και τους λοιπούς ενδιαφερομένους. Αλλά ναι, συμφωνούμε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τώρα, όσον αφορά διορθωτικού σκέλους, βάσει της ανάλυσης της Κομισιόν, δεν υπάρχει υπήρχαν λόγοι να ξεκινήσει διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών στο παρούσα φάση, αλλά σημειώθηκε ότι αν οι χώρες έχουν υπερβολικές ανισορροπίες, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν η έκβαση της συγκεκριμένης αυτής εδώ της προηγουμένης ε, παρακολούθησης θα παίξει σημαντικό ρόλο ε, και στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τι συστάσει οι χώρε και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των υπερβολικών ανισορροπιών του. Ευχαριστώ, Άλφρεντ Τσάντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η καινοτομία παρουσιάζει αδυναμίε. Ε, κόβονται κονδύλια από την έρευνα και από την καινοτομία στι ε, χώρε. Χρειάζονται ισχυρά δημοσιονομικά στι χώρε για να προωθηθούν αυτά. Συνεπώς, ε, ε, ε, διευρύνεται το χάσμα στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο των διαφορών κρατών και στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρώπη 2020 αλλά βάζει πρόσφατης ανάλυση των συστάσεων αναχώρα από την Κομισιόν διαφαίνεται ότι οι συστάσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ανομοιόμορφες Αυτές είναι οι προφορές που προέρχονται από την Κομισιόν. Ε, η αναλογία ε, έρευνας ε, και ανάπτυξη σε σχέση με το ΑΕΠ είναι στο 2%, πολύ χαμηλότερο και από τους στόχους που έχουμε θέσει εμείς και από τους, την αναλογία που υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο. Συμφωνείτε ότι μια σύγκριση, προετοιμασία των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και το ευρωπαϊκό εξάμενο ουσιαστικά οδηγούν την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη προς την ίδια κατεύθυνση. Οι διάφορε πολιτικέ δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του χάσματο καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιλογή εργαλείων πολιτική πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε τοπικέ απαιτήσει και να εφαρμόζει συνδυασμένε πολιτικέ βάσει των τοπικών αναγκών. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μέσω των συστάσεών μας δεν θέλουμε να, δείξουμε το κεφάλαιο για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη. Αντιθέτω, πιστεύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη και γι' αυτό ε, ε, ξεκίνησε και το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά ε, θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με τις μελλοντικέ τάσεις ε, και για τις ε, δημόσιες δαπάνες. Όλες οι δημόσιες δαπάνες δεν είναι ίσες, δεν είναι ισότιμες και πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει ο, ο χαρακτήρας των δημοσίων δαπανών να ενισχυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Βάνα Μαλέτιτς. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, για τα έξι κράτη-μέλη με εξαιρετικές ανισορροπίες. Σύμφωνα με την έκθεσή σας, κάποια κράτη-μέλη έχουν ανισορροπίες, τις ίδιες ανισορροπίες όπως το 2014 και 2015 σύμφωνα με την έκθεσή σας. Και κάποιες από αυτές τις χώρες δείχνουν αδυναμίες ε, στις, ε, στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ελπίζω ότι ο λόγος γι' αυτό δεν είναι η απουσία πολιτικής βούλησης, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και θα πρέπει να τονίσουμε το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όχι το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά το πώς πρέπει να γίνει, πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο. Σκοπεύετε να αλλάξετε τη διαδικασία και αντί ειδική παρακολούθησης να προτείνετε μια καλύτερη task force που θα βελτιώσει την υλοποίηση στις χώρες αυτές, γιατί ίσως να χρειάζονται κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την Συμβουλευτική Δημοσιονομική Επιτροπή στην Ευρώπη. Θα μπορούσατε να μας δώσετε την έκθεση των δράσεων που έχουν αναλυφθεί ε, για αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία. Και η τρίτη μου ερώτηση. Έχει σχέση με τον στόχο της Ολλανδικής Προεδρίας που μίλησαν για ανταλλαγή των πρακτικών και όλοι θα θέλαμε να έχουμε καλύτερη υλοποίηση και ανταλλαγή πρακτικών. Και θα ε, μπορούσε να γίνει ανταλλαγή μελετών ε, που προετοιμάζονται σε όλα τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέτοιες μελέτες θα μπορούσαν να δημοσιευθούν, να δοθούν προς όλους ώστε να ενημερωθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δομιρόφσκης. αρκετές οι ερωτήσεις σας που σχετίζονται όμως μεταξύ τους. Καταρχήν για τις ε, υπερβολικά μεγάλες ανισορροπίες και γι' αυτό που είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα όχι μόνο του τι πρέπει να γίνει αλλά και του πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί απολύτως με αυτή την αντιμετώπιση και πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια νέα δομή την υπηρεσία υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία αποσκοπεί ακριβώς στο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. το έργο αυτής της υπηρεσίας, παρότι βρισκόμαστε ακόμη ε, στην ε, αρχή, επικεντρώνεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι ακόμη στο πλαίσιο του μνημονίου, η Κύπρος ε, ήταν μέχρι πρόσφατα σε μνημόνιο. Και παρότι επικεντρώνεται λοιπόν η υπηρεσία αυτή σε αυτές τις χώρες, είναι ανοιχτή για να παρέχει τεχνική βοήθεια προς οδήποτε κράτος μέλος που θα το ζητήσει. Παραδείγματος χάρη, Συζητάμε τώρα με την ε, Κροατία για πιθανή παροχή τεχνικής βοήθειας η οποία θα παρασχεθεί από αυτή την υπηρεσία υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Άρα δεν μιλάμε μόνο για παρακολούθηση, υπάρχουν και εργαλεία για την διευκόλυνση της επίλυσης διαρθρωτικών προβλημάτων στα κράτη-μέλη. Δεν θα ήθελα ε, να συνδέσω αυτό το θέμα με την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Επιτροπή που αναφέρεται, γιατί αυτό έχει σχέση με την ε, εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για να δώσει την ανεξάρτητη αξιολόγηση των ε, δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το σύνολο της ε, Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Επιτροπή βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο δημιουργίας της. Σχετικά με τις εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή αυτή Δημοσιονομική Επιτροπή δεν έχει αρχίσει ακόμη το έργο της, όπως σας είπα, είναι σε αρχικό στάδιο. Αλλά αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται, ευχαριστώ, θα σας δώσουμε τις σχετικές εκθέσεις και πληροφορίες. Για αυτές τις μελέτες που αναφέρατε, μελέτες που γίνονται σε διάφορα κράτη-μέλη και για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε βέλτιστες πρακτικές τις οποίες θα κοινοποιούμε. Αυτό είναι ε, κάτι που ήδη κάνουμε και είμαστε πρόθυμοι να σας δίνουμε σχετική ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους Επιτρόπους για την παρουσία τους εδώ. Οφείλω να πω ότι η διαδικασία αντιμετώπισης ε, των δημοσιονομικών ανισορροπιών με έκανε να χάσω την ισορροπία μου, γιατί λέτε ότι οι συντονισμένες πολιτικές για να στηρίξουν τις ανισορροπίες ε, και να υπάρξει ανάκαμψη. Το βασικό είναι ο συντονισμός. Αλλά τι έχουμε μετά, αυτό στη θεωρία. Έχουμε εκθέσεις αναχώρα. Πώς σχετίζονται οι εκθέσεις ξεχωριστές αναχώρα με τον συντονισμό βλέπετε τον ευρωπαϊκό πυλώνα. Κάποιες πολιτικές είναι πιο ευρωπαϊκές από ό,τι άλλες. Υπάρχουν διαφορετικές εκθέσεις, ατομικές αναχώρα και αδυνατό να καταλάβω το γενικότερο σύνολο, τη γενική εικόνα. Καταρχάς. Κατά δεύτερο, διάβασα ένα άρθρο, ένα άρθρο στο νικόνομιστ όπου γινόταν αφορά στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και τον επιχειρηματικό και οικονομικό κύκλο. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Είναι κοινή γνώση αυτό για το χρονικό σημείο στο οποίο είναι καλύτερο και βέλτιστο να επέρχονται οι μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει λοιπόν το timing των μεταρρυθμίσεων να το εξετάσετε και θα μας βοηθήσει ιδιαιτέρως. Τρίτο ερώτημα. Για τις κάτω Κλασικό παράδειγμα μη ευρωπαϊκής συμπεριφοράς λέγεται και αναφέρεται ότι έχει αποτύχει δημόσια αξιολόγηση κατά 1% οι συνεισφορές στο δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος για τις συντάξεις έχουν αυξηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο το συμπέρασμα για τις κάτω χώρες, αλλά πάση είναι σαφές το συμπέρασμα. λέει ότι ο αντίκτυπος της ε, δυνατότητας επέκτασης ε, του προβλήματος από τις κάτω χώρες τους ε, εμπορικούς της εταίρους δεν είναι αρκετά τονισμένος. Ελπίζω να εξετάσετε προσεκτικά το θέμα της, κατο... της Ολλανδίας και να προωθήσετε ευρωπαϊκές λύσεις. Ευχαριστώ. Πιέχ, πολύ γρήγορα. Να σας πω καταρχάς ότι προσπαθούμε πράγματι να έχουμε μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση ε, της διαδικασίας. Άλλωστε, θέλω να σας υπενθυμίσω την συνολική θεώρηση που έχουμε για τις μεταρρυθμίσεις, για το κόστος τους, για τη μείωση των ανισορροπιών και των ε, διαφορών και ε, την άποψή μας για τις προσπάθειες για τη σύγκληση οι οποίες είναι απαραίτητες. Για πρώτη φορά έχουμε συστάσεις σε επίπεδο ζώνης του ευρώ τον Οκτώβριο του 2015, είναι το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας και θα βελτιώσουμε αυτή την ολοκλήρωση, την ενοποιημένη προσέγγιση για το σύνολο της ε, ευρωζώνης Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας για το timing, για το συγχρονισμό, πράγματι είναι πολύ σκόπιμο. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποια φάση του κύκλου βρισκόμαστε. Έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις και στην αγορά προϊόντων και στην αγορά εργασίας. Όχι οι ίδιες και όχι παντού οι ίδιες. Πάντοτε επιδέχονται βελτιώσεων και τελειοποιήσεων. Αναρωτιέμαι όμως, Μήπως χρειάζεται νέος κύκλος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην παιδεία, στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα, σε, στην ενέργεια αλλού. Ε, αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να ε, ξεπεραστεί η κρίση και από, ε, από τη στιγμή που έχουν υιοθετηθεί οι πρώτες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί η κρίση να ε, ε, έχουμε μια θεώρηση πολύ πιο μακροπρόθεσμη. Άλλωστε, πράγματι, το μέγεθος των ε, ε, χωρών δεν πρέπει να συμβάλλει και να επηρεάζει την αξιολόγηση. Η Ολλανδία είναι χώρα που είχε τεράστιο πλεόνασμα σε παράβαση του Συμφώνου Σταθερότητας. Κύριε Νίντεμάγια, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει λιγότερο σημαντικά οικονομικά από ότι πολιτικά προβλήματα. Όταν μιλάμε για την οικονομική βιωσιμότητα πρέπει να μας απασχολήσει και το βραχυπρόθεσμο γιατί αν δεν είναι καλή η πολιτική βραχυπρόθεσμα δεν θα είναι καλύτερη και αργότερα. Δεν ισχύει και αντιστρόφως. Και εδώ αναφέρομαι σε μία μελέτη της Επιτροπής πριν από λίγα χρόνια που προσπαθούσε να αξιολογήσει το κόστος που έχει σχέση με τη γύρανση του πληθυσμού, όχι μόνο συνταξιοδοτήσεις αλλά και η υγειονομική περίθαλψη κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση εδώ γιατί αρκετές χώρες έχουν ουσιαστικά προβλήματα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και κάτι πιο θετικό τώρα. Η Επιτροπή έχει φιλόδοξα σχέδια για τη βελτίωση της ίσπραξης εσόδων και υπολογίζει δισεκατομμύρια ευρώ ε, με τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Το έχετε συμπεριλάβει αυτό και στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ε, για το μέλλον και θα υποφεληθούν όλες οι χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για την δημοσιονομική βιωσιμότητα καταρχήν. Παραμένει προτεραιότητα της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης. Και όντως αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το, ο μέσος όρος του χρέους και των ελλημάτων μειώνονται. 90% του ΑΕΠ για το χρέος και 2,2% του ΑΕΠ για το έλλειμμα και αναμένεται περαιτέρω μείωση. μειούμενη τάση λοιπόν και για το χρέος και για το έλλειμμα, παρότι δεν ισχύει αυτό για όλες τις χώρες, γιατί κάποιες χώρες συνεχίζουν να έχουν υπερβολικό έλλειμμα και πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Και υπάρχουν και χώρες με πολύ ψηλό δημόσιο χρέος που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Αλλά συνολικά σημειώνουμε πρόοδο διατηρώντας ουδέτερη δημοσιονομική στάση. Δηλαδή αυτή η βελτίωση δεν προέρχεται από συμπληρωματικά μέτρα προσαρμογής, αλλά από βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Αναφέρεται το θέμα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Όταν συζητούσαμε την βιωσιμότητα, οικονομική βιωσιμότητα δεν μπορεί να μην, να είναι απαραίτητο συστατικό και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και δεδομένης της γύρανσης του πληθυσμού το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ένα από τα βασικά σημεία που μας απασχολούν και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε αρκετές χώρες εξετάζουμε τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Τώρα, για, τη για τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ίσπραξης ε, φορολογικών εσόδων. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται εντατικά με το θέμα αυτό, με προτάσεις για φορολογική διαφάνεια, για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών, υποβάλλονται προτάσεις ε, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς ε, κερδών στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του G20 προγράμματα δράσης για το ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση της απάτης στο ΦΠΑ και τα μέτρα αυτά, εάν εγκριθούν και υλοποιηθούν σωστά, θα βελτιώσουν τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. ακολουθούμε μια συνετή προσέγγιση. Δεν ε, θεωρούμε ότι έχουμε ήδη διαθέσιμα αυτά τα έσοδα τα οποία αναμένουμε μελλοντικά, αλλά εάν δούμε ότι όντως υπάρχει πραγματική πρόοδος ε, και αν συμφωνούν τα κράτη-μέλη και υπάρξουν και αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις, θεωρούμε ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση και στη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως τελευταία ομιλήτρια να κάνω μία πιο γενική ερώτηση σε δύο τμήματα. Πρώτον, όταν το Ευρωκοινοβούλιο συνέβαλε στην εκπόνηση της διαδικασίας ε, τη μακροοικονομικών ανεσορροπιών, ε, είχε την ιδέα ότι στην οικονομική συζήτηση και στη χάραξη των διαδικασιών θα προσθέταμε μία νέα διάσταση. που θα ε, προσέδιδε αυτή τη συζήτηση των υπερβολικών ανισορροπιών. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας πείτε τι δίδαγμα αποκομίσατε από όλη αυτή τη διαδικασία του MIP, σε τι χρησιμεύει, για, τι επιτρέπει να εντοπίσουμε, πώς επιτρέπει να εντοπίσουμε καλύτερα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε ε, σε σχέση με, με αυτή τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών. Και επίσης πρώτη φορά φέτος ε, αναφέρεται ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συστάσεις εντός Ευρωζώνης ε, Στι επόμενε εβδομάδε λοιπόν αυτά τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν πώ θα συντονιστούν, πώ θα συνδυαστούν μεταξύ του, και εσεί πώ θα λάβετε υπόψη τι ε, συστάσει και τα διδάγματα που αποκομίζετε από αυτή την εφαρμογή τη διαδικασία τη ΕΜΕΠΗ φέτο, ε, όταν θα συντάσετε τι συστάσεις αναχώρα. Λαμβάνοντα υπόψη και όλα αυτά που είπε ο επίτροπο ο κ. Μοσκοβισή όσον αφορά την ποιότητα των δημοσίων δαπανών και την αναγκαιότητα αξιολόγηση του κατά πόσο αναγκαίες ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και οποιασδήποτε άλλε κρίσεις μπορεί να κάνει κανείς ε, επί της φύση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προτείνονται πρώτα απ' όλα, κατά πόσο είναι ωφέλιμη διαδικασία μακροοικονομικών ενισορροπιών και πώς μπορεί να βελτιωθεί, να αναφέρω τρία στοιχεία. Πρώτον, είναι ο μόνος ε, τρόπος που έχουμε ε, για να συζητήσουμε το σύνολο του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους. Επίσης είναι ένα αντικατάστατο εργαλείο για να συζητήσουμε τη σχετική ανταγωνιστικότητα των κρατών και τρίτον ε, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για να συζητήσουμε για τα τρέχοντα πλεονάσματα. Όσον αφορά τις συστάσεις για την Ευρωζώνη, πρόκειται για μια καινοτομία, κάτι καινούριο. Η πεποίθηση μου είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ε, για να αποφύγουμε τα προβλήματα, για παράδειγμα με τους μισθούς, θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τις διαγνώσεις και στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πέραν αυτού φυσικά τίθεται ένα ερώτημα κατά πόσο αυτή η διαδικασία είναι ακριβής, δυσδυτική, αποτελεσματική. Πιστέψτε με, εμείς ε, αυτό επιθυμούμε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά όλο και περισσότερο και η βελτίωση των τελευταίων ετών με την εισαγωγή των συστάσεων για την Ευρωζώνη, με τη μείωση των κατηγοριών, με όλες αυτές τις διαδικασίες θα θέλουμε να επιτέλεσει το ρόλο της ε, και να θεωρηθεί από τις εθνικές αρχές ως κάτι δικό τους. Ε, ώστε να γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική και όλο και πιο σημαντική. Ε, αυτός που ήταν ο σκοπός ουσιαστικά αρχικά της ε, διαδικασίας ε, υπερβολικών ανισορροπιών. Πρόεδρο ευχαριστούμε. Υπήρξε πολύ επικοδομητική αυτή η συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ αυτή η ανταλλαγή απόψεων επί των οικονομικών. Να ευχαριστήσω τους αντιπρόεδρους, τον Αντιπρόεδρο κύριο Ντομπρόφσκης και τον Επιτρόπο κύριο Μοσκοβισή και τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε το διάλογο. Και τώρα δίνω το έδρα στον Σάντερ Έχουμε μια ανακοίνωση, ανακοίνωση και θα δούμε και το επόμενο σημείο της της διάταξης. Καλησπέρα συναδελφοί. Όπως φαίνεται έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες δεν έχω ακόμα δει. Um, uh- έχουμε κάποιες ανακοινώσεις του Προέδρου λοιπόν όσον αφορά τη συνάντηση των συντονιστών της 22ης Μαρτίου 1 για την οικονομική διακυβέρνηση συμφωνήθηκε η απόψινή συνάντηση έκτακτη συνάντηση με τον Επίτροπο στο πλαίσιο της έκθεσης budget και εκών για την Ευρωζώνη και ε, συμφωνήθηκε να καλέσουμε και τους Υπουργούς Οικονομικών ε, της Ευρωζώνης σε μια έκτακτη συνάντηση που θα λάβει η χώρα 11 Ιουλίου. Δεύτερη ανακοίνωση για τις αναφορές και τις προτάσεις ψηφίσματος. Οι συντονιστές συμφώνησαν επίσης να ασχοληθούν με αυτές τις αναφορές ε, και τις προτάσεις μέσω γραπτής διαβούλευση Δεν ελήφθη καμία ένσταση μέχρι την προθεσμία που ήταν την 5η 7 Απριλίου. Προ... Θα ε, υιοθετήσουμε λοιπόν το προετοινόμενο εδώ και για τα δύο θέματα. Τρίτον, για την Κίνα. Ελήφθη απόφαση αλλαγή του τίτλου της ε, ακρόασης που πρόκειται να λάβει η χώρα και ο τίτλος θα έχει ω εξή μακροοικονομικές, δημοσιονομικές, ε, χρηματοπιστωτικές ε, ε, και νομισματικές επιπτώσεις της κατάστασης στην Κίνα. Τέταρτη ανακοίνωση αφορά μια συμφωνία για μια μελλοντική αταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χίλ θα λάβει χώρα σε μια κοινή συνάντηση με την Γιούρη 20 Απριλίου και η Επιτροπή Τάξη επίσης έχει προσκληθεί. Θα εστιαστούμε στο δημόσιο CBCR. Και τελευταία ανακοίνωση για τα ζητήματα της Ομάδας Εργασίας Τραπεζικής Ένωσης. Συμφωνήθηκε να διοργανωθεί μια συνάντηση. Ε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τη σύνδεση με την κυρία ε, Κιόνι Χινούη και με την Επιτροπή. Η συνάντηση αυτή θα εξετάσει την ετήσια έκθεση Υπερτραπεζικής Ένωση του 2015. Η συνάντηση λοιπόν θα πρέπει να εξετάσει επί ζητήματα κρατικών ενισχύσεων και BRD. Και μια τελευταία ανακοίνωση. Όσον αφορά τα μέλη της ΕΚΟΝ, η ομάδα EFDD ανακοίνωσε τις ακόλουθες, τις ακόλουθες τη ε, εντός της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Θα έχουμε ως παλιό και νέο συναδέλφο την κυρία Μπέτριξ Φωνστόρχ που θα αντικαταστήσει την κυρία Νταϊαν Τζέιμς ως ε, τακτικό μέλος. Η κυρία Νταϊαν Τζέιμς θα γίνει αναπληρωματικό μέλος. Όπως γνωρίζετε η Μπέτριξ Φωνστόρχ άλλαξε ομάδες, δεν είναι πλέον ε, μέλος του ECR αλλά είναι πλέον μέλος του EFDD. Έτσι περνάμε στο επόμενο σημείο, την ε, έκθεση του κυρίου Μπαγιέ σχέση με τους κανόνες κατά των πρακτικών φοροαποφυγής. Έχετε το λόγο κύριε Συγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερω από το μήνυμα το οποίο μα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι βασίστηκε σε δικέ μα προτάσει για να διατυπώσει φιλόδοξε προτάσει προ μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Αυτή η δέσμη μέτρων που προτείνει ο επίτροπο ε, κ. Ε, Μοσκοβισή μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική καμπή και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα αντισταθεί στις πιέσει των πολυεθνικών και ορισμένων κρατών μελών και τα τελευταία σκάνδαλα με τα έγγραφα του Παναμά μας δείχνουν πόσο επίγον είναι να ε, λάβουμε μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ, η ε, επιθετική, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός του ΟΣΑ οδηγεί σε απώλειες ε, 100 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίω. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 4 και 10% των συνολικών εσόδων από τη φορολογία των εταιριών και σημαντικές απώλειε εσόδων για τα κράτη, η οποία περιορίζει την ικανότητά του να επενδύουν για την πρόθεση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχεια και την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων υγεία για όλου και για την ε, ε, ασφάλεια των χωρών. Η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς ε, και μια συντονισμένη προσέγγιση για τα φορολογικά συστήματα θα είναι ε, απαραίτητη. Προβλέπουμε με τα μέτρα αυτά να πληρώνουν οι εταιρείε ε, τους φόρους τους εκεί όπου ε, δημιουργούνται τα έσοδά τους. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι η, εγκατάσταση, ποια είναι η χώρα εγκατάστασης μιας πολυεθνικής. Γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές οργανώνονται ώστε να μεταφέρουν τα έσοδα, τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους χωρίς να έχουν πληρώσει καθόλου φόρους στις χώρες στις οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους. Έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο στην, ε, ενδομιλικές συναλλαγές Ζητάμε επίσης ε, να καταρτιστεί ε, μια μαύρη λίστα, μια αυστηρή λίστα με, αυστηρ... με φορολογικούς παραδείσους ε, που δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές φορολογικές καταστάσεις ζητάμε 10% και όχι 30% το ποσοστό που ορίζεται για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή ε, Επίση, ένα άλλο θέμα είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνία που χρησιμοποιούνται από τι ε, εταιρείε για να μεταφέρουν τι δαπάνε του ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία ε, σε χώρε όπου του βολεύει για φορολογικού λόγου. Επίση, υπάρχει η ρήτρα του switch over της προοδευτικής μεταφοράς. Θέλουμε να υπάρχει ένα, τελικά ένα δίκαιο σύστημα φορολόγησης ε, των εταιριών σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να έχουμε ε, σωστές συνθήκες ανταγωνισμού, γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι δυσμενής προς όλους. Ε, η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τον, τη φορολόγηση των εταιριών θα πρέπει ε, ε, να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο για να φορολογούνται οι εταιρείε δίκαια για τα κέρδη τα οποία υλοποιούν στα κράτη-μέλη. Είναι πολλά τα στοιχεία. Ξέρω ότι οι πολυεθνικές έχουν σημαντικά, σημαντικούς πόρους και μπορούν με το lobbying να ε, αντιταχθούν στα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε. Σχετικά πρόσφατα, στο πλαίσιο της έκθεσης ε, για τη φορολογία 1, δείξαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση και είμαστε και πάλι φιλόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα μας υποστηρίξει η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κ. Μάιερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχήν, θέλω να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής. Είναι μια καλή και εφικτή πρόταση ε, που μπαίνει προς την κατεύθυνση του προγράμματος ε, του ΟΣΑ, του BPS. και ελπίζουμε ότι θα συζητηθεί σύντομα ε, το θέμα της ε, κοινή ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιριών. Είναι μια αρκετά λογική πρόταση και ως και όδης θα προσπαθήσω να εξετάσω αν ε, υπάρχει πεδίο βελτιώσεων σε κάποιους τομείς. Το σχέδιο έκθεση νομίζω ότι θα μα δώσει πηγή έμπνευση για αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Καλό θα είναι να συμπεριλάβουμε και κάποια άλλα θέματα. Παραδείγματο χάρη, κάποιου νέου ορισμού και Κάποιες διατάξεις επίσης πρέπει να τροποποιηθούν όσον αφορά τους υβριδικούς σχηματισμούς κλπ. Δίνουμε γνωμοδότηση προς το Συμβούλιο και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εφικτές προτάσεις που θα μπορούν να θεωρηθούν αιτιολογημένες και θα μπορέσουν να είναι υλοποιήσιμες για να αυξήσουμε και την αξιοπιστία μας έναντι του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντερμάιερ. Εκ μέρους της ομάδας ECR έχω εγώ το λόγο και θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή. Θέλουμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί για να καταπολεμήσουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό αυτό είναι πολιτική προτεραιότητα σήμερα περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αποτελεί αυτό δική μου πεποίθηση αλλά και πεποίθηση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και του κόμματος οποίο, στο οποίο ανήκω. Ο ΣΑΑ προσπαθεί να ορίσει ε, κανόνες που θα ισχύουν παγκοσμίως για να παρεμποδίσουμε την μείωση της φορολογικής βάσης και την απώλεια ε, δυνατότητας φορολόγησης των κερδών. Χαίρομαι διότι τα κράτη-μέλη θέλουν να πάρουν τα μέτρα από το BEPS, από την ε, μεταφορά των κερδών, την πρόταση αυτή του ΩΣΑ. Προτείνουμε όμως να γίνει βήμα παραπάνω, πέρα από το πλαίσιο αυτό. Μιλούμε για μέτρα τα οποία ξεπερνούν αυτό το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας διεθνώς. Τα μισά μέτρα δεν βρίσκονται καν μέσα στο σχέδιο δράσης BEPS του ε, όσα. Θέλουμε να επιτεθούμε κατά μέτωπο στην αφοραποφυγή. Με το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μόλις τώρα είχαμε ένα νομισματικό διάλογο και μιλήσαμε με τους επιτρόπους. Σήμερα, σε περίοδο χαμηλής αναπτύξης και υψηλών ποσοστών ανεργίας, πάρα πολλά κράτη έχουν δυσκολίες με την ανταγωνιστικότητά τους. Άρα το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε όσο να το περισσότερες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, ήμουν σκιώδης εισηγητής για το Ταμείο Επενδύσεων του Γιούγκερ. Και ασχοληθήκαμε ακριβώς με αυτό το θέμα, πώς θα έρθουν περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Και αυτό το οποίο συζητούμε εδώ είναι μέτρα με πολύ μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής, τα οποία δύνανται να επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δύνανται βέβαια είναι η λέξη κλειδί. Ίσως φέρουν κυρίως διότι οι υπόλοιπε χώρες του κόσμου δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το το οποίο επιθυμούμε ε, εμείς, θα είναι κρίμα τελικά να πυροβολήσουμε τους εαυτούς μας στο πόδι, να ε, μπούμε σε ένα κυνήγι ε, που δεν θα φέρει αποτελέσματα και τελικά να μειώσουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη και τελικά να πλήξουμε τα νοικοκυριά, τις οικογένειες τα, σε εισοδήματα. Η φοροδιαφυγή και η φόρο αποφυγή είναι όντως πράγματα φρικτά. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις σε πλήρη συμβατότητα με τα γεγονότα και τα πραγματικά στοιχεία. Είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι δεν έχει γίνει αξιολόγηση αντικτύπου. Και αν υπάρχει ένα θέμα πάνω στο οποίο χρειαζόμαστε αξιολόγηση αντικτύπου είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν χρειάζεται αξιολόγηση αντικτύπου γιατί υπάρχει το σχέδιο δράσης του ΟΣΑ για ε, την ε, φορολογία εξόδου κατά τη μεταφορά των κερδών. Μιλούμε όμως για μέτρα που δεν είναι ε, σε αυτό το σχέδιο δράσης μόνο Επομένως θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτό το οποίο όμω με ενοχλεί περισσότερο, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση με τους σκιώδεις συζητητές είναι ε, το ενδεχόμενο να υπάρχει κρυφή ατζέντα. Ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσως είναι μια ατζέντα των μεγαλύτερων κρατών μελών εναντίον των πιο αδύναμων των ισχυρών σε σχέση με τα ε, πιο αδύναμα κρατημέλη ή με τα πιο μικρά. Είναι μέτρα που θα έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, ο περιορισμός των επιτοκίων, δηλαδή του ποσοστού των επιτοκίων που είναι φορο, που επιλέξιμα για φοροαπαλλαγές κτλ. Αυτό θα αποδυναμώσει τις πιο αδύναμες χώρες που θα έρθουν σε, ε, ε, δεν θα είναι πια ανταγωνιστικές εναντί άλλων χωρών με χαμηλά επιτόκια ούτως ή άλλως. Και τελικά οι φορολογούμενοι π.χ. της Πορτογαλίας μπορεί να μεταφέρουν την έδρα τους σε πιο ισχυρές φορολογικά χώρες όπως είναι η Γερμανία π.χ. Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε ε, περισσότερα προβλήματα. Θα έπρεπε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να αναπτυχθούν περισσότερο. Αλλά εδώ είναι το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι ισχυρές χώρες γίνονται ισχυρότερες και οι αδύναμες γίνονται πιο αδύναμες τελικά. Επαναλαμβάνω ότι αποτάσσομαι δελειρά τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Όμως να ε, μεριμνούμε και για την κοινωνική δικαιοσύνη, κυρίως για τα πιο αδύναμα κράτη-μέλη, να μην τα αποδυναμώσουμε παραπάνω. Και τώρα θα, ε, εκ μέρους του ECR παρακαλώ. Merci, ο Ενρίκε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω στα γαλλικά τον εισηγητή για την ημιτρική του γλώσσα, παρόλο που είναι Βέλγος, μητρική του γλώσσα τα γαλλικά. Όμως θα ήθελα να μιλήσω στη δική μου γλώσσα λακωνικά για να ευχαριστήσω ε, τους διερμηνείς ε, για την παρουσία τους ε, εδώ ε, και την υπομονή του στο πρόσωπό μου. Στα ισπανικά λοιπόν θα μιλήσω. Κοίταξτε, είναι αργά και θα είμαι σύντομος και για να είμαι σύντομος πρέπει να είμαι σκληρός και γι' αυτό θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Μας ενδιαφέρει και μας αρέσει η προσπάθεια που κατέβαλε ο εισηγητής. Στη δική μου πολιτική ομάδα θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε στενά την ισορροπία μεταξύ πιο πραγμάτων. Πρώτον, της δυνατότητας να ξεπεράσουμε το πλαίσιο του ΩΣΑ και να πάμε ακόμα πιο πέρα χωρίς από την άλλη να επιφέρουμε πλήγμα στην ευρωπαϊκή οικονομία και στη δυνατότητά της να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και στο επιχειρήν βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής να είναι καθησυχασμένος σε σχέση με τη δική μου πολιτική ομάδα. Εμείς θα πιέσουμε όσο θα δω περισσότερο για τις απαιτήσει και για τις βελτιώσεις ακόμα και των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ίδιος ο ΣΑ. Τώρα για τα τεχνικά, γιατί 10% εδώ, γιατί 30% εκεί. Ε, καλό θα ήταν ο εισηγητής στις διαπραγματεύσεις που επίκενται και στις συμβιβαστικές λύσεις και ούτω καθεξής να τεκμηριώσει τα τεχνικά στοιχεία ε, για τα οποία ε, ε, επιδεικνύει ιδιαίτερη φιλοδοξία. Θέλει από το 30% να φτάσει στο 10% και ούτε καν στο 15% να μας το τεκμηριώσει. Πρέπει να διαβουλεύετε με εμάς γιατί είμαστε κοινοβούλιο εδώ γιατί αυτό είναι συμπεγνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, ωστόσο οφείλει να διαβουλευτεί με εμάς, γιατί εμείς είμαστε οι πραγματικοί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Ε, όχι άμεση η δημοκρατία. Εμείς έχουμε εκλεγεί άμεσα εδώ και να μην ξεχάσουμε τα έγγραφα του Παναμά, αλλά και να τα ξεχάσουμε θα βγουν άλλα έγγραφα από άλλη χώρα και μετά άλλα και άλλα και άλλα. Έχει αρχίσει λοιπόν ο κόσμος να ε, αναρωτιέται και να είναι νόμιμα όλα αυτά και να είναι και νομότυπα. Μήπως τώρα πλέον έχουν ξεκάθαρα περάσει στη σφαίρα του ανήθικου. Ζητούμε λοιπόν από τον εισηγητή να πάει όσο πιο μακριά μπορεί, να εμβαθύνει όσο το περισσότερο. Αν όχι στα τεχνικά, τουλάχιστον στα θεμελιώδη ζητήματα. Κάτι πρέπει να πει, τουλάχιστον για τους φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η Ισπανία έχει την μεγάλη τύχη να ε, ε, συνορεύει με δύο, την Ανδόρα και το Γιβραλτάρ, για να μην πω ότι και το Μονακό είναι ε, πολύ κοντά. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι διμερείς συμφωνίες που έχουν όλες οι χώρες οι οποίες έχουν κοπιάσει να ε, υπογράψουν αυτές τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες πολύ συχνά είναι τα παραθυράκια για να διευκολυνθεί η φόρο αποφυγή θα πρέπει να έχουμε όραμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και τις υπεράκτιες εταιρείε. Να δώσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής στην νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει όμως μία ενιαία πολυμερή συμφωνία και όχι ένα σωρό διμερείς συμφωνίες με τους φορολογικούς παράδεισους. Έτσι θα έχουμε fair play και θα αποδυναμωθούν οι πιο αδύναμοι και θα αποφευχθούν οι καταχρήσεις των λιγότερο αδυνάμων. Όλα αυτά να γίνουν λογικά. Ναι, να μην διαλύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινή ευρωπαϊκή σύγκληση και εστίαση έναντι αυτού του βδελίγματος θα έλεγα γιατί τελικά ε, το φορολογικό αυτό σύστημα είναι ανήθικο. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία. Και αν κινηθεί προς τα εκεί ο εισηγητής θα τύχει πλήρους υποστήριξης από την πολιτική μου ομάδα. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ, ο κύριος Δεμάση. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο εισηγητή για την πληρέστατη πρόταση του. Δεν θέλω να σας πω όλες μου τις απόψεις για τα διαρροές των εγγράφων του Παναμά, αλλά πιστεύω ότι το σκάνδαλο δεν είναι η συμπεριφορά του Μωσεκ Φωσέκα, αλλά η διαρκής ε, ανικανότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Μιλάμε για φόρο αποφυγή, αλλά και για εγκληματικές δραστηριότητες, για χρηματοδότηση τρομοκρατίας, για ξέπλυμα χρήματος. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον Παναμά ή μόνο για τα κράτη-μέλη. Μιλάμε για χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, που δεν συμμετέχουν πλήρως στην ανταλλαγή πληροφοριών, που χρησιμοποιούν ε, κάποιες πολιτείες όπως το Delaware για το, ε, ως φορολογικούς παραδείσους και στη Γερμανία, στη δική μου χώρα υπάρχουν κάποια σημεία κάποια μέρη που είναι πιο συμφέροντα ακόμη και από τον Παναμά λόγω ανεπαρκού ε, εφαρμογή της νομοθεσίας ε, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Λοιπόν, ε, για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής ε, πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να αντιμετωπίσουμε τι ελλείψει επενδύσεων, ε, δημοσίων επενδύσεων ε, στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να επανακινήσουμε την οικονομία. Πιστεύω ότι η έκθεση αποτελεί βασική βελτίωση σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν και μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλά στοιχεία και εκτιμάμε ιδιαίτερα τι προσθήκε του εισηγητού όσον αφορά τη μείωση από 30% στο 10% του επιτοκίου. Θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε με ε, μία ρήτρα που θα ορίζει απαλλαγή των επιτοκίων ε, από τους όρους βάση ε, του κύκλου εργασιών. Θα θέλαμε ένα απόλυτο κατόφλιο 25% φόρο σε σχέση με τα πολύ χαλαρά ποσοστά του 40% που προβλέπει η Κομισιόν και καλό θα ήταν να εφαρμοστεί αυτό στο μεγαλύτερο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τρίτων μας αρέσει ε, το ότι έχει συμπεριληφθεί η εμπορία αγαθών ε, στις υπηρεσίες για τους κανόνες και η μεταφορά κερδών ε, μπορεί να γίνει με έτοιμες μεταφοράς σε σχέση με τον Κίτσο όταν αξιολογείται κατά πόσο χρησιμοποιούνται θηγατρικές διαφορά αποφυγή τέταρτων η αποκρίση για τις ασυμφωνίες ε, υβριδικών σε τρίτες χώρες ε, μας αρέσει. Πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με μια λύση που απλά να μην ευνοεί τις τρίτες χώρες. Τώρα θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ε, σε τρία σημεία. Έχουμε επιφυλάξει για τα καθεστώτα φορολογία για τι ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την προσέγγιση βάσει του συνδέσμου ε, δεν φαίνεται να έχουν αποτελέσματα. Το έχει πει και η Γερμανία το ίδιο στις ομάδες εργασίας. Τα παραδοσιακά εργαλεία όπως η φοροαπολεγή των επενδύσεων ε, έχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις και μετά όσον αφορά τους περιορισμούς των επιτοκίων θέλουμε να κάνουμε το ίδιο στο πραγματικό εισόδημα και μετά για τους κανόνες CFC. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση Ευχαριστώ πολύ. Thank you. To conclude uh, for the Greens. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζωλή, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκ για την ε, πρόταση έκθεσή του. Είναι πολύ καλή η πρότασή του και σε πολλά σημεία βελτιώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, τον ευχαριστώ για την ε, συνολική του προσέγγιση και εδώ και πολλές εβδομάδες συνεργαζόμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Η ομάδα των Πρασίνων υποστηρίζει τις περισσότερες τροπολογίες. Παραδείγματο χάρη για την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Ε, συμφωνούμε με τον ορισμό που πρέπει να δοθεί. Όσον αφορά ε, ε, την έκπτωση των ε, τόκων. Συμφωνούμε με την πρόταση να φτάσει στο 10%. Θα θέλαμε όμως μια διατύπωση που θα επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια μεταξύ ομίλων, που συχνά είναι αντικείμενο χειρισμών. Τέλος, ε, συμφωνώ με τα, το σημείο που αφορά τα patent boxes για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, που είναι μια φορολογική μάστιγα και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μέχρι τον Ιούνιο μια πρόταση και με βάση τη διαδικασία της συναπόφασης να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Ο, ο έχει ήδη επισημάνει ότι ε, τα patent boxes δεν είναι εργαλείο βελτίωσης ε, της έρευνας ε, και των επενδύσεων. Πρέπει σιγά σιγά μέχρι το 2020 να εκλείψουν και να απαγορευτούν. Ελπίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση και όλα αυτά τα σημεία θα συνεχίσουμε τα συζητάμε στις συνεδριάσεις μεταξύ σκιωδών εισηγητών και ελπίζω στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας όπως μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζολή. Επομένως σας μιλήσουμε και για τις προθεσμίες. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 15 15 Απριλίου 12 το μεσημέρι. 23 Μαΐου θα εξεταστούν οι τροπολογίες, θα ψηφιστεί στις 24 Μαΐου στην Επιτροπή Οίκων και στην Ολομέλεια θα φτάσει την, τον Ιούνιο. Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν. Κύριε Σιγητά, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Χαίρομαι που θα έχω τη δυνατότητα να συνεργαστώ και στη συνέχεια με τους ε, σκιώδεις εισηγητές μου. Εξαιρετικά, λέει ο Πρόεδρος, οπότε κλείνουμε και τη σημερινή συνεδρίαση, εκτός αν υπάρχει κάτι στα διάφορα που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας. Καλό σας βράδυ.